Μπορούμε να ξαναρχίσουμε. Έχουμε λοιπόν ε, την ακρόαση σήμερα για την προσβασιμότητα στις μεταφορές και τη σύνδεσιμότητα, τις σχετικές προκλήσεις στο χώρο της Βαλτικής. Έχουμε τρεις εμπειρογνώμονες μάλλον τρία πάνελ. Οι εμπειρογνωμένε θα μας μιλήσουν στο πρώτο πάνελ ε, για τις υποδομές στην Ανατολική Ευρώπη. Το δεύτερο πάνελ θα αναφερθεί στο πρόβλημα της ανάπτυξης υποδομών και της απουσίας ε, ε, της συνδεσιμότητας και τον αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία των πολιτών. Και τρίτον, συνέπειες, το τρίτο πάνελ, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες και ανταγωνιστικότητα. Το αργότερο θα τελειώσουμε στις 6.30. Έχουμε αρκετή ώρα λοιπόν μπροστά μας. Αλλά όπως βλέπω δεν ήταν τόσο μεγάλη, μεγάλο το ενδιαφέρον των συναδέλφων της Επιτροπής. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Δίνω λοιπόν καταρχάς για 6 λεπτά στον κύριο Τελ Τάλις Λινκάιτς, επικεφαλής της ε, γραμματείας ειδικής, της ειδικής πρωτοβουλίας για την ε, Βαλτική, ΒΑΣΑΜΠ, το λόγο. Θα μας μιλήσει για την προσβασιμότητα, για τις προκλήσεις προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας στη Βαλτική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Με μεγάλη χαρά έρχομαι σήμερα ενώπιόν σας και ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση να σας παρουσιάσω ε, τις προκλήσεις. Η Βάστα, η οργάνωση που εκπροσωπώ, είναι μια συνεργασία υπουργών αρμόδιων για, την, για τον χωρικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Πρόκειται για μια οργάνωση η οποία εδώ και 20 χρόνια παρακολουθεί τις εξελίξεις και προάγει την συνεργασία και την κινητικότητα στη Βαλτική. Ζητήματα ευρείας κλίμακος προσβασιμότητας στη Βαλτική έχουν να κάνουν περισσότερο με, την, με τις εδαφικές δομές ε, παρά με τις μεταφορές. Όπως ε, η Υπουργική Βάσαφ φέτος όρισε, ε, διαπίστωσε, έχουμε ζήτημα και γεωφυσικής προσβασιμότητας, μεγάλες αποστάσεις, μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις, διαφορετικές διαφορετικοί τρόποι μεταφορών και σημαντικές διαφορές ως προς την ε, πυκνότητα του πληθυσμού απαιτούν ε, την ε, συντήρηση των δημοσίων υποδομών, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει με επαρκή αποτελεσματικότητα. Η βελτίωση λοιπόν των δημοσίων δικτύων βελτιώνει όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη, ταυτόχρονα εξασφαλίζει συνδεσιμότητα στις μεγάλες αποστάσεις και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η ολοκλήρωση προς ανατολικά και κεντρικά και βόρεια εδάφη προς, την, προς τα τμήματα της κεντρικής Ευρώπης. Με βάση τις αξιολογήσεις των ειδικών, μόνο η, Ανατολική, η Δυτική Πολωνία και η Γερμανία στο σύνολό τους έχουν μέσο πρόθεσμο, αλλά πάντως όχι κεντρικό δυναμικό προσβασιμότητας ε, οδικής. Μέσω των σιδηροδρόμων η συνδεσιμότητα είναι καλύτερη από ότι η οδική σε σχέση με τη Γερμανία, τη Σουηδία και τη Δανία. Ωστόσο είναι εντυπωσιακό ότι είναι χειρότερη σε σχέση με την νότια Πολωνία, τη Λιθουανία και την Εσθονία. Οι ενέργειες μεταφορές εξασφαλίζουν ε, την κύρια διασύνδεση με την ε, κεντρική Ευρώπη, αλλά έχει οικονομική επιβάρυνση και δυσκολίες σε σχέση με ε, απεργίες όπως η σημερινή της Λουφτχάνσα, κυκλώνες και άλλα προβλήματα. Και δεν μπορεί να αποτελέσει τη λύση για τη μεταφορά φορτίων σε μεγάλη κλίμακα. Έχουμε βελτιώσει, ε, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο, την προσβασιμότητα για τις ανατολικές και τις δυτικές χώρες της Βαλτικής τελευταία δεκαετία. Οι ενέργειες διασυνδέσεις είναι η μόνη θετική βελτίωση που βλέπουμε για την ε, περιφέρεια της Βαλτικής, εκτός από κάποιες καινούριες γραμμές boat. οι διασυνδέσεις έχουν βελτιωθεί για ορισμένα σημεία της Φινλανδίας, της Πολωνίας αλλά και της Σουηδίας, αλλά όχι για όλη την περιοχή της ε, Βαλτικής και βρισκόμαστε ακόμη σε επίπεδο χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ολόκληρη την περιοχή μας. Δυστυχώς το δυναμικό της προσβασιμότητας με σιδηροδρόμους είναι σαφώς χαμηλότερο από το μέσο όρο της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις χώρες της Βαλτικής πλην της Γερμανίας. Υπάρχουν ελλείψεις σε επιμελητιακές ε, υποδομές, προσβασιμότητα δηλαδή στους μεγάλους θερματικούς σταθμούς, δυνατότητα πρόσβασης για τα καταναλωτικά αγαθά, καθυστερήσεις ε, για τις επιχειρήσεις. Και αυτό όλο συνεπάγεται υψηλότερο κόστος για τους τοπικούς παραγωγούς και υψηλές τιμές για τους καταναλωτές μας. Συνεπάγεται δε μειονέκτημα ως προς την ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Οι ειδικοί με την ερευνά τους αποδεικνύουν μια καθαρή και γραμμική ε, σχέση ως προς το δυναμικό προσβασιμότητας και τις οικονομικές επιδόσεις μιας περιφέρειας. Το βλέπετε σε αυτή τη διαφάνεια. Η δε Ανατολική Ευρώπη δεν έχει τις καλύτερες επιδόσεις διαφάνεια. Η Βάσαμπ επίσης έχει αναθέσει μία ε, μελέτη για την αξιολόγηση σε σχέση με τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις στην περιοχή των ε, διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και καταλήγει η έκθεση στο συμπέρασμα, η μελέτη στο συμπέρασμα ότι μπορεί να οδηγήσει σημαντική βελτίωση στην περιοχή. Λείπουν όμως κάποιοι σύνδεσμοι και παραμένουν αρκετά σημεία συμφόρησης. Επίσης καταλήγει η μελέτη αυτή ότι οι πόροι χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών δεν αρκούν για τη χρηματοδότηση όλων των προβλεφθέντων έργων η περιφερειακή συνεργασία μπορεί να στηρίξει τις εθνικές πρωτοβουλίες αλλά και τις, ε, τα έργα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ώστε να καταστήσουν πιο προσβάσιμα και βέβαια θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία στο τομέα αυτών. Αυτό κάνει η Βάσαφ. Οι Υπουργοί της Βάσαφ ε, το Σεπτέμβριο φέτος υπεγράμμισαν τη σημασία των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών για την ε, περιφερειακή ανάπτυξη και ιδιαίτερα υποστήριξαν την ανάπτυξη και υποστήριξη πράσινων διαδρόμων ε, μεταφορών και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με τα περιφερειακά δίκτυα μεταφορών των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ώστε να προαχθεί η εδαφική συνοχή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ θερμά, λέει ο Πρόεδρος, κυρίως γιατί κρατήσατε με τόση ακρίβεια το χρόνο. Σας ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ σαφή όσα μας είπατε και τώρα δίνω το λόγο για 6 λεπτά στον κύριο Γιάσο Σλάχτα από την ε, Σχολή Οικονομικών Επιστημών της Βαρσοβίας, εδαφική προσβασιμότητα εν ώψη του έργου ΕΣΠΟΝ ΕΤ 2050. Έχετε το λόγο κύριε Σλάχτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Είχα την τύχη τα τελευταία τέσσερα χρόνια να πάρω μέρος σε ένα έργο project το οποίο ονομαζόταν ε, European Territory Project 2015 ε, ε, αν μιλάμε για το θέμα της ε, προσβασιμότητας, θα πρέπει να πούμε ότι ε, η Ευρώπη είναι διαφορετική στα διάφορα μέρη της. Εδώ έχουμε το περίφημο πεντάγωνο, υπάρχουν διάφορες μητροπόλεις, ε, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης δεν είναι εύκολα προσβάσιμο. Και αν κοιτάξετε για να δείτε τις αλλαγές που επήλθαν τις τελευταίες δεκαετίες και μέχρι το και θα επέλθουμε στο 2051, θα εντυπωσιαστείτε, για δέστε σε αυτό το χάρτη, το πώς αλλάζει η Ευρώπη, για δέστε. Βλέπετε ότι η κεντρική Ευρώπη κατακτήθηκε τα έδαφος, ε, ε, ε, μάλλον είναι η κερδισμένη, το κερδισμένο ενώ τα άλλα μέρη είναι τα χαμένα. Αν λάβετε υπόψη σας την εσωτερική προσβασιμότητα, δηλαδή αν λάβετε υπόψη, υπόψη σας την πρόσβαση στις περιφερειακές πρωτεύουσες, βλέπετε λαμβάνοντα υπόψη τι υδροδρομικέ μεταφορέ και τι οδικέ μεταφορέ, θα διαπιστώσετε ότι η κατάσταση είναι μάλλον λυπηρή. Ε, στην Πολωνία ιδιαίτερα, στην Ανατολική Πολωνία, όπου ο χώρος ε, για ε, μεταφοράς ξεπερνάει τις τρεις ώρες από τη μία άκρη ως την άλλη. Προβληματική λοιπόν και προβληματικό και το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο. Ας επανέλθουμε τώρα στο πρόγραμμα ΕΣΠΟΝ υπάρχουν τρία σενάρια για το 2050. Το πρώτο αφορά την προώθηση των ε, σφαιρικών ε, των παγκόσμιων πόλεων της Ευρώπης. Βλέπετε ότι τα περισσότερα γίνονται μέσα στο πεντάγωνο, πολλά εκτός αυτού του πενταγώνου. Υπάρχει και ένα δεύτερο σενάριο. Αυτό αφορά ένα δίκτυο ε, πόλεων και την προώθησή του. Βλέπετε ότι είναι πιο εξισορροπημένο αυτό το σενάριο. Και υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο που αφορά την προώθηση των αγροτικών και περιφερειακών ε, ε, περιφερειών που έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Είναι εξισορροπημένο αλλά λιγότερο αποτελεσματικό από την άποψη στην οικονομική. Οι δικές μας ε, προτάσεις μέχρι το 2050 είναι οι κάτωθοι. Καταρχάς θα έχει σχέση ε, με το στόχο μας που είναι η πολυκεντρικότητα και το άνοιγμα της Ευρώπης. Θα πρέπει να προωθήσουμε τη σύνδεση με τις όμορες χώρες, με την Ανατολική Ευρώπη αλλά και με τη Βόρειο Αφρική. Θα πρέπει να προωθήσουμε μάλλον θα πρέπει να επιτρέψουμε την ε, ανάπτυξη, την τόπια ανάπτυξη. Σε πολλές περιπτώσεις ε, δεν δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Ε, θα πρέπει να, υπάρχει μια, να υποστηρίξουμε μια εξισορροπημένη αστική δομή και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη βιωσιμότητα των φυσικών πόρων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα εδώ, αν πραγματικά θέλουμε να ανοίξουμε τις ευρωπαϊκές αγορές στην, ε, στον ανταγωνισμό και να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα θα πρέπει να έχουμε καλύτερη σύνδεση. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ολοκλήρωση των δικτύων τηλεπικοινωνιών και μεταφορών και να ανοίξουν παγκόσμιες πύλες όχι μόνο στην κεντρική Ευρώπη αλλά και στις νέες χώρες μέλη. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν ευφυή ενεργειακά δίκτυα τα οποία θα παρέχουν πρόσβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όταν ναι, μιλάμε για την προώθηση της ανάπτυξης με σώμορες χώρες θα πρέπει να συνδέσουμε τα δίκτυα της Κεντρικής Ευρώπης με αυτά των όμορων χωρών και να προωθήσουμε την εδαφική ανάπτυξη διακρατικά, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας ε, για το θέμα των ε, ε, διαφορών μεταξύ των χωρών και της τοπικής ανάπτυξης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να έχουμε επαρκείς υποδομές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο γιατί πολλές πολλές πολλές περιφέρειες συνεχίζουν να μην καρπούνται τα πλεονεκτήματα που έχουν στη διάθεσή τους. Εδώ έχετε τα δίκτυα δίκτυα της Ευρώπης και εύκολα μπορείτε να δείτε ότι η χειρότερη κατάσταση παρατηρείται στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Καρπαθία Οδός θα μπορούσε να έχει περιθώρια για να αυξήσει την προσβασιμότητα. Δεν είναι σημαντικός ο άξονας Ανατολής αλλά και Βοράς και Ανώτου. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία που μπορείτε, στα οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από το www.espon.eu και ET2050. Επιτέλους ευχαριστώ αυτούς που συνέβαλαν στο να διαμορφώσω αυτή την ομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου. Και τώρα περνάμε στην επόμενη ομιλία πάλι 6 λεπτά για το Ματίας Γιούρεκ της UNEP. Προστορνή γραμματεία της Καρπαθικής Συμβάσεως της Βιέννης θα μας μιλήσει για τη βελτιστοποίηση των υποδομών μεταφορών με την ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορών φορτίων και επιβατών. Έχετε το λόγο. Thank you also very much for the very kind invitation, in particular to Mr. Tomos Poreba, for giving us the opportunity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 ασκείται ιδιαίτερη πίεση στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει κίνδυνο στη συνδεσιμότητα. Το σημαντικό είναι ε, να έχουμε συνδεσιμότητα αλλά και αηφορία και προσβασιμότητα. Οι χώρες ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις προκλήσεις δεν μιλούμε μόνο για την πίεση που ασκείται στο περιβάλλον, μιλούμε και για τον τουρισμό. Πάρα πολλές περιοχές μέσα στα Καρπάθια δεν είναι καθόλου προσβάσιμες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε ήπια κινητικότητα και ανάπτυξη του τουρισμού. Οι χώρες έχουν επιτύχει να διαπραγματευτούν ένα πρωτόκολλο, ένα κείμενο νομικός δεσμευτικό, αυτό το υπέγραψαν, το υιοθέτησαν οι Υπουργοί της περιοχής των Καρπαθίων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είναι ένα σημαντικό νομικό εργαλείο για την αηφόρο μεταφορά επιβατών και εμπορεύματος. Έρχεται να συμπληρώσει τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την σχετική νομοθεσία. Έχουμε την προσέγγιση της προφύλαξης σε βασικούς ε, τομείς και αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ ευρύ το πλαίσιο αυτό και οι χώρες συμφωνούν να εστιάσουν τον ενδιαφέρον τους σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, οδικές, σιδηροδρομικές ε, μεταφορές, αλλά και μεταφορές μέσω των πλωτών οδών. Δεν θέλουμε μόνο να μειώσουμε τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και να βρούμε καλύτερους τρόπους για να το πετύχουμε αυτό, αλλά θέλουμε και πολυτροπικές συνδέσεις και καλύτερη διαλειτουργικότητα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αναλάβει διάφορα έργα ΑΚΚ Project για την αποκατάσταση της οικολογικής συνδεσιμότητας μεταξύ της Βιέννης και της Μπρατισλάβα. Πολλές δραστηριότητες βιομηχανικές αλλά και που άπτονται άλλων πεδίων. Συνεργαζόμαστε με διάφορες επιχειρήσεις για να χτίσουμε γέφυρες και να αποκατασταθεί αυτός ο οικολογικός διάδρομος σε διευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόσβαση στις ορεινές περιοχές. Αυτή είναι η προσέγγιση μας και τη χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λύσεις ήπιας κινητικότητα. Στην ιστοσελίδα θα δείτε ότι οι εταίροι στο έργο αυτό έχουν καταλήξει σε πολύ καλές ε, πρακτικές για τον τρόπο με τον οποίο θα προωθηθεί η αηφόρος κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Καρπαθίων. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον. Τρεις είναι. Καταρχάς, να στηρίξουμε τις χώρες να επικυρώσουν και να υλοποιήσουν το πρωτόκολλο μεταφορών. Είναι ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό εργαλείο. Το θέμα του τελευταίου μιλίου, δηλαδή πώς θα έχουν καλύτερη προσβασιμότητα οι κάτοικοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της περιοχής των Καρπαθίων. Και τρίτον, κάτι που στηρίζει η τσεχική ε, Προεδρία της Σύμβασης των Καρπαθίων είναι το θέμα των πράσινων υποδομών. Πώς η βιοποικιλότητα μπορεί να ε, βρεθεί στο επίκεντρο των διαφόρων πολιτικών στους διάφορους τομείς έτσι ώστε να υπάρχουν ωφέλη για τους πολίτες. Στο πλαίσιο λοιπόν της σύμβασης των ε, Καρπαθίων θέλουμε οι πράσινες υποδομές να συμβάλλουν στη συζήτηση που γίνεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί όπου χαράσεται η πολιτική αλλά και επί τόπου όταν μιλούμε για την υλοποίηση της εκάστοτε πολιτικής. Με αυτές τις γραμμές λοιπόν, με αυτά τα λόγια θα ολοκληρώσω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι μας αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κρατημέλη και αυτό είναι καλό, ότι δηλαδή η Σύμβαση των Καρπαθίων είναι ένας μηχανισμός, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο σε περιφερειακό επίπεδο και μας βοηθάει να εφαρμόσουμε διάφορες πολιτικές και για τις μεταφορές και υπέρ της βιοπικιλότητας. Άρα, σε ό,τι μας αφορά, ε, το σημαντικό είναι να ακολουθήσουμε την αρχή της προφύλαξης. Η εφόρος ανάπτυξη δεν έχει μόνο να κάνει ε, με, την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και με την προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων μέσω του παραδείγματος της σύμβασης των Καρπαθίων μπορεί ε, να φανεί ε, πολύ καλύτερα πώς βρίσκεται το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ όλων αυτών των πυλώνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν και οι τρεις ε, παρουσιάσεις. Πριν περάσουμε στη συζήτηση θα ήθελα να καλωσορίσω δύο ομάδες επισκεπτών. τον Ντομινίκ Ρικέ, η πρώτη, μια αντιπροσωπεία 12 επισκεπτών από την Εθνική Ομοσπονδία των Οδικών Μεταφορών προερχόμενοι μάλιστα από διάφορες πόλεις της Γαλλίας. Καλώς ήρθατε. Και η δεύτερη ομάδα είναι εκπαιδευόμενοι διερμηνείς. 15 τον αριθμό. Καλώς ήρθατε και εσείς στην Επιτροπή μας. Ποιος θέλει το λόγο τώρα? Κύριος Φαντανκάμπ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Διαπιστώνω κάποιες διαφορές στις ε, παρουσιάσεις. Είδαμε μια success story για προκλήσεις ε, που αντιμετωπίστηκαν, ενώ η άλλη παρουσίαση μιλούσε περισσότερο για τις προκλήσεις που παραμένουν. Αυτό που δεν πολύ κατάλαβα όμως και απευθύνω το ερώτημα προς τους τρεις ομιλητές είναι το εάν το πρόβλημά σας είναι κυρίως οικονομικό ή έχει να κάνει με ιδέες, υποδομές, αδειοδοτήσεις. Ερωτώ λοιπόν εάν μπορείτε να μου δώσετε κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί πολύ συχνά αποδίδουμε τα προβλήματα στην έλλειψη χρημάτων. Όμως ε, η συνεργασία μεταξύ των ε, βαλτικών κρατών ε, ίσως να μην έχει προχωρήσει όπως θα έπρεπε και να υπάρχουν και κάποια κενά στη χάραξη πολιτικής. Επίσης σε σχέση με την Ουκρανία, η οποία είναι μέρος των έργων για τη συνδεσιμότητα, θα ήθελα να ρωτήσω η κατάσταση που επικρατεί, τι επιπτώσεις έχει, συνεχίζεται σαν λογικοί άνθρωποι που είστε ή όλα τα πράγματα έχουν πια πολιτικοποιηθεί τόσο που σταματάει το, σχέδιο. Αυτό ήταν οι ερωτήσει μου. Ποιο άλλο θέλει το λόγο. Η κυρία Μάισνερ. Όχι, δεν ήταν η κυρία Μάισνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φανκάμπ, με, με προλάβατε. Οι δύο παρουσιάσεις δείχνουν κάποιες αρνητικές εικόνες ε, και πρέπει να συμφωνήσω εγώ, μια και προχωράμε από την περιοχή Πορκαπάτσε. Έχουμε βέβαια ένα σοβαρό λόγο για τον οποίο έχουμε καθυστερήσει τόσο στην ανάπτυξη των δικτύων, ότι βρισκόμαστε πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα για τόσα χρόνια, ενώ από την άλλη πλευρά η Γερμανία μπορούσε να προχωρήσει και να αναπτυχθεί. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να αναγνωριστεί ότι τις καθυστερήσεις της η Ανατολική έχει καλύψει αρκετά γρήγορα στην περίοδο που έχει μεσολαβήσει από το 90 και μετά. Θα ήθελα να αναφερθώ δε στα προβλήματα της προσβασιμότητας που πρέπει να ε, επιληθούν. Λέγεται ότι έχουν μείνει πολλά προβλήματα ακόμα. Ναι, αλλά μην ξεχνάμε και όσα έχουν ε, αντιμετωπιστεί. Υπάρχουν πολλά έργα, έργα υποδομών, ο κύριος Γιούρεκ αναφέρθηκε σε κάποια ζητήματα που μένουν ακόμη εκκρεμοί, αλλά τόσα έχουν γίνει. Δεν θέλω να περάσει αυτή η ακρόαση σαν ε, ένας, ε, μια ευκαιρία για πολιτική εκμετάλλευση και καταγγελία του ότι κανένας δεν αναλαμβάνει μέτρα εδώ. Δεν ισχύει αυτό. Ο καθένας θέλει να περάσουν τα μέτρα, να εγκριθούν, να εφαρμοστούν μέσα σε μια πενταετία και βέβαια δυστυχώς ο χρόνος δεν φτάνει. Για την Βοηβότικα Πότκα Πάτσε αναφερθήκατε σε διάφορες διασυνδέσεις και ανάγκη και διασυνδέσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν τα προβλήματα. Αναπτύσσετε το οδικό δίκτυο, αλλά αναπτύσσετε και το σιδηροδρομικό δίκαιο. Πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά. Και υπάρχουν έργα που χρηματοδοτούνται χάρη σε διαγωνισμού, σε προκηρύξεις. Αλλά μερικές φορές δεν είναι ακριβώς σαφές ποιες δραστηριότητες προάγονται και πού πάνε τα χρήματα. Πάντως ήταν χρήσιμο και ενδιαφέρον το ότι αναφερθήκατε στο ζήτημα αυτό, γιατί η περιοχή αυτή, η Fort έχει ζητήματα. Έχει ζητήματα προσβασιμότητα, ε, σύνδεσιμότητα, αλλά δεν θέλω να δοθεί εντύπωση ότι δεν γίνεται και τίποτα. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ και Ζήνε Μάισνερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση προ όλου του ομιλητέ για τον κύριο Λινκάιτ, Καταρχά τον πρώτο ομιλητή που μας είπε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες. Κοιτάξτε, αυτό είναι πάγιο πρόβλημα στον τομέα των μεταφορών. Η Επίτροπος Μπούλτς ήταν σήμερα εδώ και μας μίλησε για τις ε, προτάσεις ε, για το μέσον συνδέοντας την Ευρώπη. Τι μπορείτε λοιπόν να προβλέψετε εσείς από τη δική σας την πλευρά, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί και τι είδους βελτίωση στη χρηματοδότηση θα μπορούσατε να προβλέψετε ανάλογα με το τι μπορούν να στήσουν τα κράτη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκραπίνη έχει το λόγο. Μία συγκεκριμένη ερώτηση σε ό,τι αφορά τις τρεις προτεραιότητες που παρουσιάσετε για το μέλλον. Αναφέρω ότι θέλετε να υποστηρίξετε τις χώρες που θέλουν να εφαρμόσουν αυτού του είδους τα έργα. Το θέμα είναι πώς. Κάθε φορά που έχουμε ακροάσεις όλοι έρχονται και μας λένε τι πρέπει να γίνει κανείς, δεν μας λέει πώς πρέπει να γίνει. Με κάθε ειλικρίνεια δεν κατάλαβα καλά τις προτεραιότητές σας. Εγώ ζω στη Ρουμανία και αυτή η σύμβαση των Καρπαθίων με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υπάρχει όμως και η στρατηγική του δει. Εγώ διετέλεσα υπουργό και πρέπει να σας πω ότι η στρατηγική αυτή δεν απέδωσε πάρα πολύ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιο είναι ο στόχος αυτής της σύμβαση των Καρπαθίων, γιατί εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ισορροπίας. Η ανάπτυξη των υποδομών, όπως είπατε, ασκεί πίεση στο περιβάλλον. Ωραία. Πώς θα επιρρήσουμε την εξίσωση αυτή έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή υποδομή αλλά να μπορούμε να προφυλάξουμε και το περιβάλλον. Εγώ θέλω να ακούσω κάποιον ειδικό. Να μην μιλάμε μόνο για τις ε, πολιτικές, να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές λύσεις που θα μπορούσαμε να βρούμε. Τόμας Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής και τον πρόεδρο που οργάνωσαν την ε, ακρόαση αυτή για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την ε, προσβασιμότητα για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Κατά την άποψή μας πρόκειται για μια περιφέρεια που ακόμα δεν έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη σε όλα αυτά τα επενδυτικά προγράμματα που είμαι σίγουρος ότι ε, αν κάποια στιγμή θα γίνονται θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτή η περιοχή και θα συνέβαλαν παράλληλα στην βασική λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότητα ευκαιριών. Αυτή είναι η λογική μας. Θέλουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτυχθούν με έναν εξισορροπημένο τρόπο μεταξύ τους. Η κατάσταση είναι τέτοια που στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη σε ό,τι αφορά το θέμα της προσβασιμότητας της επικοινωνίας ένα θέμα τόσο σημαντικό από όλες τις απόψεις, η περιοχή αυτή δεν λαμβάνεται παρκώς υπόψη. Πολύ συχνά γιατί υπάρχει απουσία πολιτικής βούλησης από πλευράς των κυβερνήσεων για τις συγκεκριμένες χώρες. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Περάσω τώρα στο δεύτερο. Σήμερα συζητάμε για το τι θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε η προσβασιμότητα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα ήταν δυνατόν να βελτιώσουμε τις επικοινωνίες μεταξύ της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και των υπόλοιπων μερών της Ευρώπης, έτσι ώστε οι κάτοικοι της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Βουλγαρίας να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι χάρη σε αυτούς τους δρόμους, τις οδούς τραχίας κυκλοφορίας ή χάρη στην γρήγορη μεταφορά των εμπορευμάτων κατάφεραν να λύσουν μερικά από τα προβλήματα που καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν. Εγώ δεν τρέφω ελάχιστη αμφιβολία για το γεγονός ότι η Καρπαθία Οδός που στην Πολωνία την ονομάζουμε S19 θα συμβάλλει σε μια γοργή ανάπτυξη, θα δημιουργήσει δηλαδή καλύτερες ευκαιρίες μεταξύ της σχετικής και Ανατολικής Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Εάν κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος, θα καταφέρουμε να επιλύσουμε πολλά από τα προβλήματα με τα οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι σήμερα, ενώ άλλα θα καταφέρουμε να τα αποφύγουμε εντελώ. Δεν θα ήθελα η ακρόαση αυτή να γίνει ένα, μια σκηνή όπου συγκεντρώνονται πολιτικοί διαξεφισμοί. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν υπεγράφει στην Πολωνία μια συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών το χρόνο που βρίσκονται κατά μήκο της καρπαθιας Οδού και σε αυτή τη συμφωνία δηλωνόταν η πρόθεση στο άμεσο μέλλον να δημιουργηθεί αυτός ο δρόμος. Δυστυχώς πολλά χρόνια πέρασαν και όπως έλεγε ο κύριος Βουκατσεύσκ, όντως ε, δημιουργείται, ε, κατασκευάζεται ένα μέρος της Καρπαθίας Οδού. Το, το υπόλοιπος δρόμος όμως που θα πρέπει να φτάσει μέχρι τα σύνορα με τη Λιθουανία και μετά μέχρι τη Σλοβακία δεν κατασκευάζεται και δεν υπάρχει και καμία προοπτική κατασκευής του. Δίχως άλλο, ούτε το 15 δεν θα ξεκινήσουμε. Με λίγα λόγια, απαιτείται πολιτική βούληση. Επιτρέψτε μου να καταλήξω κύριε Πρόεδρε. Εάν είχε υπάρξει στο παρελθόν η πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί αυτό το έργο, θα περούσαμε σε μια ιδιαίτερα προχωρημένη φάση. Δυστυχώς υπάρχει το συμπληρωματικό μέρος, αλλά δεν υπάρχει το βασικό μέρος. Εν συντομία, διακόπτει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε λίγο. Οι ομιλητέ μα είχαν από 6 λεπτά ο καθένα και πρέπει να δώσουν και απαντήσει. Ε, δεν είναι δυνατόν εσεί να μιλάτε περισσότερο από αυτού, α του σεβαστούμε. Σα παρακαλώ σύντομα. Καλά. Τρία λεπτά. Τρία λεπτά δώστε μου. Το τελευταίο μου σχόλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε σήμερα προβούμε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά έτσι ώστε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δέσουμε κάποια προτεραιότητα σε αυτό το δρόμο. Έτσι ώστε να, να κατασκευαστεί το συντομότερο δυνατόν. Εντάξει. Λοιπόν, το μέγιστο είναι τρία λεπτά. Δεν είναι υποχρεωτικό να τα εξαντλήσετε βέβαια. Απλώς να μπορέσουν και οι άλλοι να μιλήσουν. Τρία έτσι, όχι δύο. Πολύ γενναιόδωρος είστε, Πρόεδρε, αφού μας δίνετε τρία και όχι δύο λεπτά. Λοιπόν, τίτλος της ακρόασης είναι «Συνδεσιμότητα, ε, πρόσβασιμότητα στην κεντρική Ανατολική Ευρώπη». Δεν είναι μόνο τα Καρπάθια. Το κατάλαβα αυτό. Έχουμε μια νέα πολιτική μεταφορών στην Ευρώπη, τα TEN-T, διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Έχουμε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο δίκτυο και έχουμε τον εισηγητή της σχετικής έκθεσης εδώ μαζί μας. Νομίζω λοιπόν ότι πράγματι η Ευρώπη έχει κάνει κάτι για όλα αυτά τα πράγματα, για τη συνδεσιμότητα και την προσβασιμότητα όλων των περιφερειών στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ευρώπης. Πρέπει όμως και εμείς να κάνουμε κάτι. Έχει έρθει η στιγμή κατά την οποία μέσω της συνεργασίας των κρατών μελών της εκάστοτε περιφέρειας μπορούμε πράγματι να κάνουμε κάτι. Έχουμε το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη, έχουμε την πολιτική συνοχής, έχουμε το σχέδιο το επενδυτικό, έχουμε το, το Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Υπάρχουν κονδύλια δηλαδή. Με τη συνεργασία των χωρών μελών μπορούμε να υλοποιήσουμε τα διάφορα έργα που θα συνδέσουν τις χώρες μας. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό και τι ξέρετε για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Κλόντια Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά χρήσιμη και εξαιρετικά σημαντική και χαίρομαι διότι δίνουμε έμφαση στις επενδύσεις και στην υποδομή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις επί των έργων υποδομών στην συγκεκριμένη περιοχή. Με το πρόγραμμα TEN-T τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών καλούμαστε να αποφασίσουμε επί συγκεκριμένου προγράμματος και πρέπει να αποφασίσουμε και να εγκρίνουμε συγκεκριμένες προτάσεις έτσι ώστε να είναι πιο απρόσκοπτη η σύνδεση με τις ανατολικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να προβλέψουμε και άμεσες συνδέσεις με τη Δυτική Ευρώπη. <clears throat> και αυτό το σημείο σχολιάστηκε το πρωί που είχαμε συζήτηση με την Επίτροπο κυρία Μπούλτσο. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συνδέσεις και με το εξωτερικό, με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι θέμα υποδομών, είναι θέμα οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, οι οποίες θα ανθίσουν με τις μεταφορές. Και γι' αυτό θέλουμε συγκεκριμένες προτάσεις και εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου μπορούμε να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις στις χώρες μας, να εξηγήσουμε τι θα πει διάδρομος με την ευρωπαϊκή έννοια του όρου, με την έννοια που, δίδεται σε αυτή τη λέξη από το TENTI, έτσι ώστε η Ευρώπη να συνδέεται με τις υπόλοιπες χώρες, τον υπόλοιπο κόσμο, τη Ρωσία και γιατί όχι να μην φτάσει και μέχρι την Κίνα η σύνδεσή της. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα αυτό, οφείλουμε να το υλοποιήσουμε, να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, ιδέες για να γίνει αυτός ο διάδρομος πρόσβασης προς την Ανατολή πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ναι, βεβαίω είναι πολύ καλό να κάνουμε αυτέ τι διασυνδέσει, αλλά θέλω να επισημάνω ότι εδώ πέρα έχουμε, έχουν περάσει τόσα χρόνια που είμαστε ενωμένοι Ευρώπη και θα πρέπει να βρούμε λύσει για τα κράτη τη Ανατολική και τη ε, περιοχή τη Βαλτική. Η σιδηρόδρομη είναι μία, ε, ένα μπάλωμα μια κουβέρτα όλων μπαλώματα και ακριβώς στα σύνορα των κρατών βρίσκονται τα προβλήματα και οι συμφορήσεις. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα λοιπόν. Τα προβλήματα που έχουμε, τα κράτη-μέλη λένε δεν θέλουμε να τα λύσουμε. Άρα την κύρια, την κύρια ευθύνη πρέπει να την αποδώσουμε στα κράτη-μέλη για το ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Ναι. Αλλά ξέρουμε και τις ελλείψεις. Και για την Πολωνία ιδιαίτερως. Η Πολωνία ήθελε να μεταφέρει 1,2 δις χρηματοδότησης που είχαν προβλεφθεί για τους υδροδρόμους σε έργα για τις οδικές μεταφορές. Έχω ξέρω πολλά έργα, 30, 40 και εσείς ασφαλώς και περισσότερα θα ξέρετε, επενδύσεων στην Πολωνία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτές τις διασυνδέσεις. Αυτό συνισχύει και για τα άλλα κράτη. Προτείνουμε λοιπόν, αλλά δυστυχώς το Συμβούλιο δεν δέχθηκε και η Επιτροπή, το κομμάτι από τα σύνορα μέχρι την προσοχή σιδηροδρομικό κόμβο να ενισχυθεί κατά 85% από τα διαρθρωτικά ταμεία, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Τώρα πρέπει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αυτοί οι κόμβοι οι οποίοι έχουν καταστραφεί και έχουν μείνει στην καταστραφή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υποστηρίζονται. Και επίσης, θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, θα ήθελα να σας ρωτήσω πού εντοπίζετε τις κύριες ελλείψεις, τα κύρια ελλείμματα ώστε και εμείς να δώσουμε την ε, ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά. Πρέπει να ενισχυθούν λοιπόν τα σημεία συμφόρησης και διάσπαστο συνδέσμου. Έχετε λοιπόν τώρα καθένα σας από τρία λεπτά για να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω εν συντομία. Η παρουσίασή μου πράγματι τόνισε τις ευκαιρίες κυρίως. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στο περιβάλλον είναι σημαντικός. Αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι πράγματι υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά υπάρχει και αντίκτυπο στο περιβάλλον και γι' αυτό πρέπει να εντοπίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να τις διαδώσουμε. Και αυτό υπάρχει, δεν αρχίζουμε εκ του μηδενός δηλαδή. Έχουμε με τη Σύμβαση του Καρπαθίου στρατηγικά έργα, στηρίζουμε τις χώρες ε, τις κυβερνήσεις για να υλοποιήσουν αυτά τα έργα και τα, στα έργα αυτά εμπλέκεται και η οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, εμπλέκεται ο ιδιωτικός τομέας, εμπλέκονται ε, διάφοροι φορείς που έχουν εμπειρία για το πώς, για παράδειγμα, χτίζεται μία πράσινη γέφυρα, ε, πώς το οικολογικό σχέδιο γίνεται αναπόσπαστο μέρος του γενικότερου σχεδίου. Θέλουμε να εντοπίσουμε τις καλές πρακτικές και να τις αναπαράγουμε σε άλλες περιφερειές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για την περιοχή των Καρπαθίων, αλλά ισχύει και για άλλες περιοχές όπως είναι η περιοχή των Άλπαιων. Οι Αυστριακοί, για παράδειγμα, στις Αυστριακές Άλπεις έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία ε, σε σχέση με ε, την πρόσβαση στο βουντό, τις πράσινες μεταφορές, τις πράσινες υποδομές και έχουμε εντοπίσει, ε, έχουμε καταρτήσει ένα κατάλογο εκατοντάδων καλών πρακτικών έτσι ώστε να ξέρουμε τι πρέπει να γίνει σε τεχνικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο. Έχω μαζί μου ε, μια σύνθεση όλων αυτών ε, εάν σας ενδιαφέρει. Μιλούμε λοιπόν για capacity building και αυτό είναι σημαντικό και στη Σύμβαση των Καρπαθίων θεωρούμε ότι η εφόρος ανάπτυξη επιτυχάνεται μόνο όταν έχουμε πολυτομεακή προσέγγιση και εντοπίζονται οι σύνδεσμοι, οι σύνδεσμοι με άλλα πεδία και άλλους τομείς σημαντικούς. Το νομικό εργαλείο το εκάστοτε εργαλείο πολιτικής αποφασίζεται και δημιουργείται με τη συμβολή όλων. Στο πρωτόκολλο για τις μεταφορές έχουμε στελέχη από το Υπουργείο Μεταφορών, από το Υπουργείο Τουρισμού και ούτω καθεξής. Ε, γίνεται ε, μεγάλη συζήτηση για το σωστό σημείο ισορροπίας, έτσι ώστε και να εξυπηρετούνται οι μεταφορές και να υπάρχει οικολογική ε, ισορροπία αν θέλετε, η προστασία του περιβάλλοντος. Όλα αυτά στη θεωρία είναι καλά, τα έχουμε κάνει και μπαίνουμε τώρα στην πράξη και προσπαθούμε να τα υλοποιήσουμε. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις χώρες υπ' αυτή την έννοια. Αυτό που τόνισα στο τελευταίο σημείο της παρουσίασής μου είναι το εξής. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να τονίσουμε τη σύνδεση ε, με το όλο θέμα της πράσινης υποδομής, γιατί υπήρξε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ένα θέμα στο οποίο η Ευρώπη έχει προχωρήσει αρκετά και ε, ε, κοιτούμε πώς θα το εφαρμόσουμε, τις καθαρές, τις πράσινες υποδομές στην περιφέρεια που μας ενδιαφέρει. Ε, οι μεταφορές θα πρέπει να συμβαδίζουν με την προστασία της βιοποικιλότητας. Στα Καρπάθια, λοιπόν, μετά την απόφαση των Υπουργών, ε, συζητούμε το ενδεχόμενο συνεισφοράς έτσι ώστε να υπάρχει πράσινη υποδομή. Οι μεταφορές είναι σημαντικό κομμάτι όλων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πραγματικά είναι πρόκληση να καταφέρω να απαντήσω σε τρία λεπτά σε τόσο πολύπλοκες ερωτήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσω να πω κάτι. Καταρχάς, πώς είναι, σε τι σημείο φτάσει η εξέλιξη των πραγμάτων. <clears throat> Μιλάμε για 300 χιλιόμετρα από την Βαρσονιμιτία, αλλά ο, χώρος, ο χρόνος που απαιτείται για να ε, να διασκήσει κανείς αυτή την περιοχή με το τρένο είναι 6-7 ώρες. Εμένα το τρένο μου αρέσει πολύ, αλλά μιλάμε για απαράδεκτες καταστάσεις. Μας χρειάζεται καινοτόμο σκέψης, γιατί οι περιοχές αυτές βρίσκονται κοντά στα εξωτερικά σύνορα. Και εμείς θα πρέπει να καταφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα σε αυτές τις περιοχές. Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν ορισμένα σημεία εκκρεμή. Θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που είναι πολύ κακής ποιότητας και το ότι είναι ορεινές οι περιοχές δεν είναι δικαιολογία. Ύστερα χρειαζόμαστε καλές σχέσεις με την ε, Ουκρανία θα πρέπει τα σύνορά μας να είναι πιο μικρά αυτά που είναι τώρα. Το δοκιμάσαμε με την Ρωσία. Εφαρμόσαμε ένα καθεστώς εκτός έγκεν και στέφτηκε από επιτυχία αυτή η προσπάθεια. Γιατί άραγε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια προσπάθεια και με την Ουκρανία. Μια προσπάθεια να βελτιώσουμε την υποδομή, τις υποδομές μεταξύ της Πολωνίας και της Ουκρανίας. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η πυκνότητα της κυκλοφορίας δεν είναι το μοναδικό μας μέλημα. Γιατί σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Πολωνίας είναι χαμηλή η πυκνότητα της ε, κίνησης γιατί δεν υπάρχουν καλές διασύνδεσεις. Δίχως άλλο η κίνηση θα αυξηθεί όταν επέλθουν αλλαγές. Και Χαίρομαι που τα συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. Χαίρομαι που αλλάζουν τα πράγματα. Ο δρόμος <coughs> είναι έτοιμος όταν είναι από την αρχή μέχρι το τέλος έτοιμος. Μιλήσαμε για το θέμα χαμηλής προσβασιμότητας στις περιφερειακές πρωτεύουσες και όχι μόνο στην πρωτεύουσα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ε, βελτίωση της διασύνδεσης μεταξύ των διαφόρων χωρών γιατί δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ο πιο γρήγορος τρόπος ε, για να φτάσει κανείς ε, είναι να διανύσει μια υπόσταση που θα χρειαστούν τρεις ώρες. Ο κύριος Λίνκαρ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις τόσο πολύπλοκες ερωτήσεις που μου θέσατε. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τη σειρά μου ότι θα χρειαστούν πολλές ώρες για να ε, δούμε γιατί υπάρχουν αυτά τα κενά μεταξύ της Κεντρικής Ευρώπης και της ε, Ανατολικής Ευρώπης. Θα έλεγα ότι δεν είναι, τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν και διαφορές τεχνικού χαρακτήρα που έχουν σχέση με τα, την διαλειτουργικότητα. Υπάρχουν και διαφορές στην νοοτροπία των ανθρώπων στις διάφορες χώρες και θα ήθελα να παραθέσω ένα παράδειγμα του αεροδιαδρόμου του Βαλτικού αεροδρόμου ε,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 τους ομιλητές και πάνω απ' όλα τους ομιλητές από το πρώτο πάνελ. Αλλάζουμε τώρα και περνάμε στους ομιλητές από το δεύτερο πάνελ. Άννα, Όρτιλ και Πόντο. Thank you.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 σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε λοιπόν το θέμα της ανάπτυξης των ε, υποδομών μεταφορών και της απουσίας διασυνοριακών συνδέσμων, η φωνή των περιφερειών και της κοινωνίας των πολιτών. Είμαστε ολίγοι βέβαια δυστυχώς σήμερα, αλλά μπορώ να δώσω το λόγο στους ομιλητές. Ο κύριος Όλταν Πάινα είναι ο πρώτος και πρόεδρος της ε, επαρχιακής συνελεύσεως Χάιντου Πίαρ της Ουγγαρίας. Και θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Κύριε Πάινα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, η επαρχία αυτή, η Χάιντου Μπιχάρη, είναι μια από τις ε, πολύ μικρές περιοχές στην Ανατολική Ουγγαρία. Τέταρτη όμως σε πυκνότητα πληθυσμό. Θα ήθελα να σας δώσω κάποια στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούμε τα ε, χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογουμένου σε έργα μεταφορών και τηλεπικοινωνιών. Είχαμε λοιπόν ε, την την κατασκευή τους τα τελευταία χρόνια των αυτοκινητοδρόμων M3 και M35, μεγάλες, ε, μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη κυρίων οδικών ε, αξώνων, την ανάπτυξη του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ντεμπρέτσεν, ε, ανακατασκευή πάνω από 100 σιδηροδρομικών γραμμών. Όλα αυτά βοήθησαν ιδιαίτερα στην ε, προσβασιμότητα στην περιοχή και την ανταγωνιστικότητα. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δομές. Είμαστε στα εξωτερικά σύνορα του Σέγγεν, μαζί με τη Ρουμανία, κατά τα άλλα στο κέντρο της Ευρώπης. Γεωγραφικά. Στο Ζοβοτνότ. Στο Ντέμπρετσεν που βλέπετε στα νότια και στο Χοϊντουμπίντου που είναι το σημείο το κομβικό. Το βάρας νος νόμιν είναι ένα σημείο διακλάδωσης του αυτοκινητοδρόμου μη 35. Και έχουμε και πρόσβαση για το αεροδρόμιο με τα μεγάλη ταχύτητα σιδηρόδρομο μέχρι 135 χιλιόμετρα την ώρα. Έτσι λοιπόν είναι συνδεδεμένο το Ντέμπρετσεν με τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της Ευρώπης. Έχουμε ένα μεγάλο σημείο ε, διάβασης των συνόρων. Έχουμε ένα αεροδρόμιο με επιμελητιακή βάση στο Ντέμπρετσεν και μικρότερα σημεία διασύνδεσης, η κόμβη διασυνοριακοί που διευκολύνουν τη μεταφορά προσώπων και φορτίων σιδηροδρομικούς. Παρ' όλα αυτά όμως, το δυναμικό μεταφορών μεταξύ Ρουμανίας και της δικής μας επαρχίας είναι πολύ χαμηλό. Από το 2007 στο 2013 αναπτύχθηκαν πολλές, ε, πολλά έργα υποδομών, κυρίως τα σιδηροδρομικά που σας ανέφερα νωρίτερα, Όσον αφορά τα λειτουργικά προγράμματα για τις μεταφορές, έγιναν πολλά έργα ανακαίνησης, κυρίως για τα πιο μεγάλα φορτηγά. Η εθνική υπαριθμών 4 και υπαριθμών 5 επίσης ανακαινίστηκαν, έγιναν έργα. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα. Αυτό που μπορούμε να προγράψουμε για το μέλλον είναι ότι στο τέλος ε, της ε, περίοδου αυτής της πενταετής θα πρέπει να έχουμε προσβασιμότητα για όλους τους ε, μεθοριακούς σταθμούς. Μέχρι το 2016 πιστεύουμε ότι θα πρέπει να φτάνουμε με αυτοκινητόδρομο στα ρουμανικά σύνορα, πράγμα το, πράγμα το οποίο ακόμη δεν έχουμε εξασφαλίσει. Και ακόμη και μέχρι την Ουκρανία. Περιμένουμε να είναι έτοιμος αυτοκινητόδρομος στο 2016 περαιτέρω όμως θετική εξέλιξη δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ακόμη. Η Εθνική παριθμόν 4 η οποία πρέπει να επεκταθεί, να διευρυνθεί για να γίνει όχι αυτοκινητοδρόμος, αλλά πάντως να έχει δύο λωρίδες, θα πάει μέχρι το Σλουντάνιε με τις δύο αυτές λωρίδες και πολλά από τα έργα των υποδομών χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα η επαρχία μας συνορεύει με τη Ρουμανία. Βλέπετε στο πράσινο τους μεθοριακούς σταθμούς και μέχρι το 2020 θα αναπτυχθούν και άλλοι αντίστοιχοι σταθμοί στην Ουγγρο-Ρουμανική Μεθόριο αλλά και στην Γερμανο-Ουγγρική Μεθόριο. Εφέτος το καλοκαίρι οι Ρουμανικοί μας με την Ουγγρική κυβέρνηση υπέγραψαν συμφωνία που πρόκειται να συμβάλλει στην διασύνδεση μικρών πόλεων και χωριών που βρίσκονται από τις δύο πλευρές των συνόρων αλλά που δεν έχουν μεταξύ τους συνδεσιμότητα. Τις βλέπετε στο χάρτη. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι τώρα δεν έγινε καμία δουλειά για την διασύνδεση αυτών των παραμεθόριων πόλεων και γι' αυτό υποφέρουν σε επίπεδο και οικονομικό και κοινωνικό. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βλάτισλαβ Όρτιλ τώρα από την περιοχή Ποτ Καπάτσκι θα μας μιλήσει για ένα ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι σημαντικό στοιχείο ε, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης είναι πολύ απλά η βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Και αυτό είναι επίσης αληθές για την περίπτωση της Πολωνίας. Θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι η πολιτική συζήτηση είναι αυτή που θα πρέπει να οδηγήσει στη λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Σήμερα όμως είμαστε εδώ σε αυτό το πάνελ ως ομάδα εμπειρογνωμόνων και προσπαθούμε να προβληματιστούμε για όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη της εκάστοτε περιφέρειας, της χώρας ή και ολόκληρης της Ευρώπης. Ας δούμε λίγο το χάρτη. Έχουμε τον αυτοκινητόδρομο S19, ο οποίος διασχίζει την Ανατολική Πολωνία, την Ανατολική Σλοβακία, την Ανατολική Ουγγαρία και αυτές είναι και οι πιο αδύναμες περιοχές και στην Ευρώπη και στις χώρες τους. Και γι' αυτό αυτός ο αναπτυξιακός άξονας είναι εξαιρετικά απαραίτητος και υψώνεται μία τροχοπέδη σε αυτή την ανάπτυξη και είναι τα καρπάθια όρη. Πρέπει να διασχίσουμε τα βουνά χωρίς να καταστρέψουμε το, το περιβάλλον για να συνδεθούμε καλύτερα. Μιλούμε για 700 χιλιόμετρα περίπου αυτοκινητόδρομου και μόνο τα 50 έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Είναι ένα έργο που μόλις έχει ξεκινήσει, ενώ υπάρχουν και τμήματα που δεν παρουσιάζουν συνοχή, που είναι κατατεθμημένα, που υπάρχουν κενά, που παρουσιάζουν κενά. Και αν δούμε ε, το μερίδιο που έχουμε ήδη υλοποιήσει, τα 50 χιλιόμετρα στα 700 χιλιόμετρα συνολικά οδικού δικτύου, ε, βλέπουμε ότι έχουμε κάνει μόλις το πρώτο βήμα. Θέλουμε όμως να ανοίξουμε τα Καρπάθια προς την νότια δική μας περιοχή, αλλά και να ανοίξουμε όλες αυτές τις περιφέρειες περισσότερο προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλουμε μία προσέγγιση βήμα-βήμα, σταδιακή, γιατί η οικονομική πρόκληση είναι τεράστια και δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην πρόκληση αυτή σε άμεσο χρόνο. Το πάνω κομμάτι έχει ξεκινήσει. Το κάτω κομμάτι όμως, έτσι όπως φαίνεται στο χάρτη, θα αποτελέσει την πρόκληση του μέλλοντος. Και έτσι όλα αυτά είναι απαραίτητα για να ελευθερωθεί η πόλη του Ρεζ, που είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας, να αποσυμφορηθεί, γιατί η κατάσταση είναι τραγική από πλευράς κίνησης. Έχουμε και άλλες πόλεις, Μπογουχόβα, από την οποία, είναι μια πόλη από την οποία περνούν 80.000 οχήματα κάθε μέρα. 30 ή μάλλον χιλιάδες οχήματα κάθε μέρα και σύμφωνα με τις προβλέψεις το 2030 αν δεν κάνουμε κάτι θα φτάσουμε στα 80.000 οχήματα κάθε μέρα που θα περνούν από αυτή την πόλη. Ε, κάτι το οποίο θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ε, ρήπανση θα αυξήσει ιδιαίτερο στη ρήπαση, την μόλυνση, ενώ τα επίπεδα οθορύβου ε, θα φτάσουν στα ύψη. Ήδη ισχύει αυτό στις αστικές περιοχές. Δεν μιλούμε μόνο για την πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά πρόβλημα είναι εξίσου τα, η μεγάλη χορύπαση. Θα θέλαμε λοιπόν ε, με τα επιχειρησιακά ε, προγράμματα για τις υποδομές και το περιβάλλον να ολοκληρώσουμε το πρώτο στάδιο, ενώ το δεύτερο στάδιο θα υλοποιηθεί με το ανατολικό πρόγραμμα ε, και το πρόγραμμα που έχει να κάνει με την Πολωνία και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα διάφορα ευρωπαϊκά κονδύλια είτε μέσω του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη είτε μέσω άλλων εργαλείων. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολλαπλές οι πηγές χρηματοδότησης και έχουμε τις εθνικές συμβάσεις οι οποίες θα έρθουν να δέσουν μεταξύ τους όλα αυτά τα μέσα χρηματοδότησης. Βλέπετε τις μπλε κουκίδες στην διαφάνεια, στην οθόνη. Εκεί είναι τα διάφορα αναπτυξιακά έργα που γίνονται. Επενδύσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Όλα αυτά θα γίνουν εφικτά χάρη στο νέο αυτοκινητόδρομο. Βλέπετε ότι υπάρχει συνέργεια μεταξύ των μεταφορών και των άλλων ειδών επενδύσεων και όλα αυτά θα οδηγήσουν σε κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αυτής της περιοχής και εν γέννη της χώρας. Πιστεύω ότι μπορεί όλο αυτό να λειτουργήσει ως παράδειγμα, όχι μόνο για την Πολωνία, τη δική μου χώρα, αλλά και για τις υπόλοιπες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς δηλαδή ολόκληρες χώρες ή περιοχές χωρών μπορούν να ξαναγεννηθούν μέσω του αυτοκινητόδρομου ΣΥΓΜΑ 19, εάν επιτύχουμε τις συνέργειες. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο καθηγητής Πόπο που θα μας μιλήσει για διακρατικά δίκτυα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι είμαστε ένα δίκτυο οργανώσεων που εστιάζουν την προσοχή τους στο περιβάλλον. Τα χρήματα που επαιδείονται σε έργα που θα μπορούσαν να πλήξουν το περιβάλλον. Η οργάνωσή μας εστιάζει την προσοχή της στον προγραμματισμό των, ε, στα νέα λειτουργικά προγράμματα 2014-2020. Επειδή οι περισσότεροι από εμά Συμμετείχαμε σε ομάδες εργασίας. Καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα που θα θέλαμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Πρόκειται για προκατακτικά συμπεράσματα και ενδεχομένω θα επέλθουν ορισμένε αλλαγέ. Παρ' όλα αυτά. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. σε ποια συμπεράσματα έχουμε καταλήξει. Και κοιτάξτε, το, τη διαφάνεια αυτή αφορά τις επενδύσεις, τις μεταφορές το 2014 με το 2020. Ε, ε, προσέξτε την ε, αριστερή πίτα Βλέπετε ότι έγιναν σημαντικές αλλαγές στην περιβαλλοντική πολιτική σε ό,τι αφορά τις μεταφορές. Παρ' όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι για την ώρα δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα παρόμοιο συμπέρασμα όταν δούμε την ανάλυση αναχώρα. Παρόλο που οι σιδηροδρομικές μεταφορές αποτελούν προτεραιότητα μέχρι το 2020, βλέπουμε ότι οι περισσότερες χώρες μέλη στην περιοχή μας πρωτίστως επενδύουν στις οδικές μεταφορές. Ενδεχομένως η μόνη εξαίρεση εδώ είναι η Ουγγαρία. Ακούγοντας ε, τις διάφορες παρουσιάσεις, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το επίπεδο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών πολιτικών και αυτά που έχουν υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους. Έχουμε πολιτικές που έχουν την υποστηρίξη της πλειοψηφίας, όταν δεθεί όμως το θέμα των εθνικών προγραμμάτων και το θέμα της κατανομής των πόρων συμβαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες. Αυτά είναι ευρήματα και συστάσεις με βάση τη δουλειά που κάναμε στον τομέα των μεταφορών. Δηλαδή το διαδικτυακό δίκτυο μεταφορών και άλλη διάδρομη. Λαμβάνοντας ε, λοιπόν αυτά υπόψη, οι επενδύσεις που προτείνονται για το 2014-2020 δεν ε, πληρούν, δεν είναι σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές ε, πολιτικές και τις πολιτικές μεταφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώσαμε ότι οι επενδύσεις μέχρι το 2020 δεν θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα μεταφορών της περιοχής μας. Βεβαίως γινόμαστε μάρτυρες συστηματικών παραβιάσεων των περιβαλλοντικών νόμων. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και το διαδικτυακό δίκτυο, όπου υπάρχει συστηματική παραβίαση ορισμένων κανόνων, μη συμμόρφωση. Έτσι ε, έχουν τα πράγματα στη Βουλγαρία, έτσι έχουν τα πράγματα στην Βουλγαρία και σε πολλά άλλα μέρη που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε εκτενέστερα κατά τη διάρκεια του χρόνου των ερωτήσεων. Φαίνεται ότι για την ώρα οι εθνικές κυβερνήσεις της χώρα μας λαμβάνουν υπόψη τους εκτιμήσεις των επιπτώσεων και όχι τις υπάρχουσες συνθήκες, την υπάρχουσα κατάσταση. Και φαίνεται να υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό θέμα εδώ. Στις περισσότερες χώρες το σύστημα μεταφορών δεν εξετάζεται με έναν ολιστικό τρόπο, υποδιαιρείται σε υποομάδες ο τομέας των αερομεταφορών, των χερσαίων ή των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με αυτόν τον τρόπο είναι ανεπαρκή τα κονδύλια που δίνονται. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις όλα προκαθορίζονται στα υπουργικά γραφεία και ούτε το κοινό ούτε άλλοι συμφεροντούχοι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να επηρεάσουν τα πράγματα πριν από την εφαρμογή και μετά κατά τη φα... ε, ε, ε, ε, ε πριν από την υιοθέτηση κατά τη φάση της εφαρμογής. Ευχαριστώ. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε ερωτήσεις απαντήσεις. Ποιος έχει ερώτηση ή σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές για τις παρουσιάσεις. Έχω μια γενική παρατήρηση μόνο. Η πατρίδα μου, Κεντρική Ευρώπη, Τσεχική Δημοκρατία, δεν είναι αντικείμενο της ε, σημερινής συζητήσεως μεν. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες γενικευμένες παρατηρήσεις. Είναι σημαντική λοιπόν αυτή η συζήτηση και γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί ως προς την Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, λέγοντας ότι οι διαφορές στις υποδομές των μεταφορών μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να απαλληφθούν. Πρόκειται για προϋπόθεση της συνοχής στις μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Ο κύριος Κράμερ το ανέφερε ήδη. Η υπερσυνεριακή σταθμή διασύνδεσης είναι πολύ σημαντική. Εμείς έχουμε ως, ως ε, Τσεχία πολύ καλές διασυνδέσεις με την Γερμανία, αλλά και προς Ανατολάς, με τη Σλοβακία, ξέρετε ότι ήμασταν ενωμένο κράτος, ε, ακόμη και πίσω από το σύντριμο με ένα κράτος. Ε, προς τη Σλοβακία. Παρόλα αυτά δεν είναι τόσο καλές οι διασυνδέσεις και είναι οι περιοχές της Τσεχίας που βρίσκονται στα ανατολικά μας σύνορα είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. Πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στις ε, υποδομές των μεταφορών είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα εδώ να επιβεβαιώσω ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τα διαθέσιμα κονδύλια, αλλά και ζήτημα βούλησης, πολιτικής βούλησης των κυβέρνησεων των κρατών μολών. Με αυτήν μπορούν να γίνουν οι επενδύσεις. Βέβαια έχει γίνει μια αρκετά καλή προετοιμασία των έργων μεταφορών και Πιστεύω ότι οι εντάσεις σχετικά, σημαντικές εντάσεις που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, ακόμα και σε σχέση με ε, οικολογικές ενώσεις, και αντίστοιχα πιέσεις από τις κυβερνήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρατηρήσεις ε, και για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Ντέλη. Όχι, ο κύριος Ντέλη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Είναι περίτω πιστεύω να τονίσουμε το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των περιφερειών στην υπόθεση αυτή. οι περιφέρειες είναι πολύ σημαντικές. Και γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω εδώ εκπροσώπους των περιφερειών στην ακρόασή μας. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή και βαρύτητα στις περιφέρειες. Και πρέπει και αυτές να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απαραίτητη προβλεψιμότητα, δηλαδή να μπορούν να προγραμματίζουν με βάση σταθερές, ε, σταθερά δεδομένα και να προχωρούν στα έργα που τις ενδιαφέρουν. Μαθαίνουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές προτάσεις ε, για έργα από, τον, ε, από τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Σήμερα το πρωί ακούσαμε άλλωστε και την Επίτροπο που μας μίλησε για το θέμα αυτό. Από εδώ τη συζήτηση προέκυψε ότι υπολογίζεται πως μπορούν να αντληθούν κονδύλια από το, τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. και ότι θα κρυθούν ε, τα έργα ανάλογα και με τις θέσεις εργασίας που μπορεί να δημιουργήσουν και την ποιότητά τους γενικότερα. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν αρκετές θέσεις εργασίας. Εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με την ανάγκη για υποβολή ποιοτικών προτάσεων έργων. Και αντίστοιχα βέβαια πρέπει να ελεγχθεί τι είδους κονδύλια, τι είδους απόδοση πριν αφιερώσουμε όλο το χρόνο και το χρήμα στα έργα αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι αξίζουν και αντίστοιχα να τα υποστηρίξουμε. Εδώ είναι καθοριστική σημασία στο να υπάρχουν οι κανόνες, να μην αλλάζουν συνέχεια και πρέπει να προσέξουμε να υποστηρίζονται τα έργα και από τις περιοχές αυτές για τις οποίες συζητούμε, όπως άλλωστε μας ανέφερε η Επίτροπο σήμερα το πρωί, με βάση τα ποιοτικά αυτά στοιχεία. Σας ευχαριστώ, κυρία Λουκασέφσκα. Ε, ε, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ, όλους τους εμπειρογνώμονες για τις εισηγήσεις τους. Δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Είναι σημαντικές τέτοιου είδους, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και πρέπει να εκτυλιχθούν σε, στις περιφέρειες. Στο τοπικό επίπεδο χρειάζονται επενδύσεις και εκεί γίνονται πιο ε, εύληπτες, πιο κατανοητές. Και πολύ συχνά το τοπικό επίπεδο αγνοεί ε, ποιου είδου σχεδιασμός είναι ο καλύτερος. Ε, αυτά τα οποία είπε και ο καθηγητής κ. Σλέχτε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, οι πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω είναι και οι, οι καλύτερες. Και άλλωστε η παρουσίαση για το πολωνικό αυτοκινητόδρομο ε, είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί δείχνει πόσο θα συνδέσει ο S19 τις υπόλοιπες χώρες. Περνάει από τις ανατολικές περιοχές πολλών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης ούτως ή άλλως. Και πολλοί έχουν υπογραμμίσει ότι από πλευράς υλοποίησης των μεγάλων επενδύσεων το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι πιο φυσικά, η οικονομική πόρη. Και χαίρομαι, διότι διαπιστώνω ότι στα Καρπάθια δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Υπάρχουν κονδύλια, συγκεντρώνονται κονδύλια από διάφορες πηγές χρηματοδότησης ή επένδυσης και ελπίζω ότι ε, όλα αυτά τα έργα θα επεκταθούν και σε άλλους τομείς επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τους ομιλητές από το πάνελ για τις πολύ συγκεκριμένε αναλύσεις που μας παρουσίασαν για την ε, περιοχή στην Ανατολική Πολωνία, τη Μισκομαζόρσκη, προς τη Βαλτική, Έχουμε δέκα διαδρόμους που ορίστηκαν από τελευταία θετία. Για αυτούς προβλέπεται ένα συντονιστής, ο οποίος συντονίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες ε, κυβερνητικές αρχές, των Υπουργών Μεταφορών, προσδιορίζει τις λεπτομέρειες, συνεργάζεται με τα εκάστοτε κράτη. Δεν ξέρω αν και με τη δική σας την περιοχή στην Πολωνία ε, με τις τοπικές αρχές δηλαδή ή μόνο με την κεντρική κυβέρνηση της Πολωνίας συνεργάζεται και προσδιορίζει με τον τρόπο αυτόν προτεραιότητες. Συγκεκριμένα δηλαδή ένας άξονας θα αναπτυχθεί, θα έχει εύρος, μήκος και όλα αυτά αντίστοιχο με την πιθανολογούμενη επιβάρυνσή του από μεταφορές. Έτσι λοιπόν, ο διάδρομος από την Αθήνα στην Κωνσταντζα και τη Βαλτική, περνώντας δηλαδή από τον Εύξηνο Πόντο πηγαίνει στη Βαλτική, και από εκεί αντίστοιχα από τον Εύξηνο Πόντο και την Μεσόγειο προς το βορρά είναι ένα έργο το οποίο την χάνει αυτό το συντονισμό ή εμπίπτει σε αυτό το συντονισμό. Από τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη έχουμε επενδύσει όχι μόνο στον χώρο των μεταφορών προβλέψει και το ξέρει ο κύριος Κράμερ πολύ καλά γιατί το έχουμε συζητήσει αλλά έχουμε και 11 δις ευρώ από το Ταμείο Συνοχής από τα μέσα συνοχής για τα οποία είπαμε ότι θέλουμε αυτά τα υπερσυνοριακά έργα να καλυφθούν χρηματοδοτικά. Έτσι λοιπόν έχουμε συνολικά 24 δις ευρώ επενδυτικό όγκο. Η Επίτροπος Μπόλς μάλιστα σήμερα μας καθησύχασε όλους ότι ε, με την ε, μόχλευση αυτών των εργοσίων 15 δις ε, που προβλέπεται να είναι διαθέσιμα θα μας μείνει και το ποσό που έχουμε στη θέση μας για να πούμε ότι θα μεγαλώσει. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που μας προέβλεψε. Πολύ σημαντική δήλωση. Διότι εάν θέλουμε πράγματι να αναπτυχθεί η οικονομία, να έχουμε ανάπτυξη οικονομική και θέσεις εργασίας, growth and jobs, πρέπει να ε, ενισχύσουμε τις υποδομές. Και αυτό σε κάθε περιοχή και στις περιφερειακές, για να μπορούν να πολλούνται τα προϊόντα παντού και να κυκλοφορούν. Ε, ειδικά όμως και για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουμε μια επιπλέον δυνατότητα για τις επενδύσεις στις ε, υποδομές μεταφορών από, το, από τα διαφορετικά ταμεία. Ναι, πρόεδρε, τελειώνω που να είναι. Τα οποία ποσά προβλέπονται ακριβώς για τα συγκεκριμένα αυτά κράτη. Και ναι, για 25 χρόνια μας χώριζε το συντηρούν παραπέτασμα και οι, στόχοι, περιοχές στόχου, στόχου 1 ανήκανε μόνο στη Δυτική Ευρώπη μέχρι τη διεύρυνση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολο ήταν να αναπτυχθούν τα έργα των υποδομών. Ο συντονισμός όμως αυτός είναι άκρος σημαντικός και γι' αυτό σας ρωτάω εάν έχετε την επαφή με τους συντονιστές αλλά και με τους εκάστοτε υπουργούς της κεντρικής κυβέρνησης ώστε σε συνεργασία μαζί του να αναπτύσσονται οι προτεραιότητες και να κάνετε δουλειά υπερσυνοριακή cross-border. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας. Πολύ σύντομα σας υπόσχομαι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σας και να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς κύριε Πάινα καταρχάς σε εσά απευθύνομαι. Ε, ποια είναι η άποψή σας για το εξής. Είναι δυνατή η σύνδεση της στρατηγικής των Καρπαθίων με τον αυτοκινητόδρομο των Καρπαθίων. Δεν θα μπορούσε η Καρπάθια οδός να είναι το βασικό στοιχείο της στρατηγικής. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Στρέφουμε τώρα στον κύριο Ποπόφ και σας ρωτώ το εξής. Κατά τη γνώμη σας, οι, οι περιβαλλοντικές πτυχές τις οποίες αναφερθήκατε, ποιο αντίκτυπο θα έχουν στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις προτεραιότητες ε, των μεταφορών. Δηλαδή, περιβαλλοντικές αποφάσεις σε ποιο βαθμό επηρέασαν ή επηρεάζουν τα έργα που ε, ε, επιλέγησαν. Ήταν καθοριστικό το περιβαλλοντικό σκέλος ε, στην, για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στρέφομαι προς τον Πολωνό διοικητή της περιφέρειας. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιδέα σας. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις ιδέες που μοιραστήκατε μαζί μας. Θέλω να ασκήσετε περισσότερη πίεση στην Πολωνία, ώστε να μεταφέρονται τα κονδύλια, το είπε και η Επίτροπος Μπούλτς σήμερα, δηλαδή ε, να παίρνουμε κονδύλια από το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη για να τα διοχετεύουμε σε νέα έργα τα οποία συμβαδίζουν περισσότερο με το σχέδιο ε, Juncker. Εάν η πολωνική κυβέρνηση έχει πάρει το θέμα στα σοβαρά και είναι αποφασισμένη, τότε θα υπάρξει πρόοδος. Θα το συζητήσετε με το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Πολωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα εγώ είμαι ο τελευταίο στον κατάλογο. Καταρχάς πρέπει να σημειώσω την κατάπληξή μου για το ότι οι δύο πρώτοι ομιλητέ μίλησαν μόνο για οδικού άξονες. Γιατί δεν πάμε λίγο πιο πέρα, γιατί μπορούμε βεβαίως να καλύψουμε τις ανάγκες σε οδικές μεταφορές, αλλά μπορούμε και να μειώσουμε το οδικό δίκτυο ώστε να σπρώξουμε τις μεταφορές σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Ε, στην Γερμανία, παραδείγματι, όταν έγινε η εξηγένση του άξονα μεταξύ Κάρστ και Μπέκμαν, είχαμε πολύ γρήγορα μεταφορά του ε, φορτίου, την ενίσχυση λέει, του φορτίου που μεταφερόταν από τον οδικό άξονα. Το αντίστροφο λοιπόν μπορεί να γίνει. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης, χτίζοντας μόνο νέους δρόμους ή μήπως ε, κατασκευάζοντας υποδομές ε, μεταφορών ταχείες και ε, πρακτικές Ξέρετε, όταν ήταν ε, δήμαρχος του Μίνχενο Φόγκελ, που ήταν και ο νεότερος ότι δήμαρχος, είχε πει ότι ε, το οδικό δίκτυο ε, το χτίζουμε όλο και περισσότερο, αλλά κάποια στιγμή φτάνει σε ένα σημείο κορισμού και δεν μπορούμε να το αυξήσουμε περισσότερο. Και οι ανάγκε στι μεταφορέ δεν ικανοποιούνται και άρα θα πρέπει ούτω ή άλλω να στραφούμε προς, άλλες, προς άλλους τρόπους μεταφορών. Για δε την οικονομική αποδοτικότητα υπάρχουν πολλά παραδείγματα από την Γερμανία και δε την Ανατολική όπου όλοι προσπαθούσαν, όλοι έτειναν προ την κατασκευή οδικών αξώνων και την χρήση του αυτοκινήτου. Είδαν όμω πολύ γρήγορα ότι δεν προσφέρει την οικονομική ευρωστία ε, ο τρόπος των οδικών μεταφορών μόνος του για να προχωρήσει μια χώρα. Και επίσης οι στόχοι και οι επενδύσεις, ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικές σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Έχει γίνει ανάλυση ότι 60% των κονδυλίων πάνε, μόνο, σε οδικές μεταφορές, μόνο 40% στους ιδιοδρόμους, 2% για τις υποδομές ποδηλάτων. Η Ουγγαρία μας μιλάει βασικά για τις ε, ανάγκες της σε σιδηροδρομικό δίκτυο, Και έχει μεγάλη σημασία να κοιτάξει και τις ε, μεταφορές ε, σε, με ποδήλατο. Γιατί όσο χτίζουμε βέβαια δρόμους και δίνουμε το βάρος στις οδικές μεταφορές, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτε για το περιβάλλον. Πρέπει να κοιτάξουμε άλλους τρόπους, αηφόρους τρόπους μεταφορών. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν, ιδιαίτερα για την Ουγγαρία αλλά και για τις άλλες χώρες που μεταφέρθηκαν και για την Πολωνία επίσης που μεταφέρθηκαν ενώ προβλέπονταν για την ενίσχυση του σιδηροδρομικού δικτύου στις οδικές ε, υποδομές, υπάρχει τρόπος να τα δούμε διαφορετικά, υπάρχει τρόπος να αναγνωρίσουμε ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να έχουμε καλές σιδηροδρομικές μεταφορές από ότι τα 50 χιλιόμετρα ενός αυτοκινητοδρόμου που χτίζεται εδώ και τόσα χρόνια και που τελικά δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες μας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ήταν πολύ περιορισμένο ο χρόνος μου και γι' αυτό ε, θεώρησα ότι θα μπορούσα να ε, αγγίξω και στο θέμα των ε, σιδηροδρομικών υποδομών είχαμε 5 δις για την περίοδο στο 2020 στην Ουγγαρία και έχω επικοινωνήσει με αρκετές περιφέρειες. Ο άξονας Βουδαπέστης Μίσκολς είναι πάρα πολύ σημαντικό σε παραδείγμα της για τις μεταφορές. Έχουμε και άλλες ιδέες για την ευρύτερη περιοχή της Βάρδας, της Ρουμανία και πολλά άλλα κομμάτια και διασυνοριακές διασυνδέσεις. Και στον Τέμπρετσεν επίσης έχουμε κάνει μια μελέτη σκοπιμότητας χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε, που ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να οδηγήσει στην ε, κατασκευή ενός συγκεκριμένου έργου που θα ενισχύσει το δυναμικό μας ε, των μεταφορών και θα μετατοπίσει το βάρος από τις οδικές μεταφορές. Στον Τέμπρετσεν ε, υπολογίζουμε την, την κατασκευή ενός έργου αρκετών εκατομμυρίων ευρώ σιδηροδρομικού που να διευκολύνει και τις μεταφορές μικρών αποστάσεων. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να υποστηριχθεί. Είναι στη τελευταία ανάλυση μια λύση, η οποία δεν σημαίνει απαραίτητα δίλημα και διληματικές επιλογές μεταξύ οδικών δικτύων και σιδηροδρόμων. Θέλουμε να έχουμε ένα καλό δίκτυο και πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη προχωρήσει σε πολύ καλό δρόμο. Φυσικά μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο το σιδηροδρομικό δίκαιο. Για τους ε, στόχους μας είναι στρατηγικός στόχος αυτή η φάση της ανάπτυξης να συνεχίσει ακόμη περισσότερο για την Καρπαθία οδό προς ε, Ανατολάς και Νότιο-Ανατολικά με τον αυτοκινητόδρομο με 35 για το Μίσκολς και το Κάσαου έχουμε πολύ σημαντική είναι πολύ σημαντικός ε, ε, μεθοριακός σταθμός ή μάλλον διασυνοριακή διασύνδεση και θα θέλαμε να τον υποστηρίξουμε επίσης. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Mm, oczywiście rozpocznę odpowiedź od e, Pańskiej kwestii. Ja chcę powiedzieć, że... Θα ξεκινήσω απαντώντας τα ερωτήματα που μου απευθύνατε. Έξι λεπτά τα για αυτούς που δεν είναι συνηθισμένοι στα κοινοβουλευτικά δεδομένα ε, φαίνεται ε, πραγματικά βουνό. Μου φαίνεται δύσκολο να καταφέρω να απαντήσω σε έξι λεπτά. Μιλάμε για τις ε, τους ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Υπάρχουν ορισμένε σιδηροδρομικές γραμμές ε, στη Νότια Πολωνία που δεν χρησιμοποιούνται παρκώς. Για το λόγο αυτό πολύ συχνά παραμελήθηκαν. Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε ότι υπάρχουν επενδύσεις που αφορούν τις ε, σιδηροδρομικές, ε, τις αεροπορικές και τις χερσαίες μεταφορές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις μεταφορές γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές. Την περιοχή αυτή της Πολωνίας κατοικεί το 1 τέταρτο του πολωνικού πληθυσμού. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για την περιοχή των Καρπατίων, αλλά για όλη την Ευρώπη. Μιλάμε για μια περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα, μέσα στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι επενδύσεις έχουν υποστεί μια επιβράδυνση λόγω της οικονομικής κατάστασης. Παρόλα αυτά θα ήταν αναγκαίο να επιμείνουμε. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορα στοιχεία, διάφορα δεδομένα, συμπεριλαμβάνοντα και το οικολογικό. Μιλώντας για τη Τσεχία, μιλάμε πάντοτε για δίκτυα, δεν μιλάμε για κλειστό σύστημα επικοινωνιών. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάμε πέρα από τα εθνικά και περιφερειακά μας σύνορα. Σε ό,τι αφορά τις δικέ μας υποδομέ θα έλεγα ότι πρόκειται για θετικές υποδομές. Χρειαπαιτούνται όμως 2 δισεκατομμύρια που λείπουν για να συνεχιστεί η εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Η απάντηση, η απόφαση για την οποία μίλησε η Επίτροπος είναι μια σημαντική απόφαση. Εμείς σαφώς είμαστε υπέρ του να διπραγματευτούμε περαιτέρω συμβάσεις για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο. Η κυβέρνηση όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να το ε, κινητοποιηθούν. Το θέμα είναι να μπορέσει να μπει κάποιο τέλος στο κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό αυτών των περιοχών. Κατά την άποψή μου η σημερινή συζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική και δίχως άλλο θα συμβάλλει στις μελλοντικέ εργασίες δίχως άλλο θα επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη. Βεβαίως υπό τον όρο ότι θα εφαρμοστούν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ποπόφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να απαντήσω στις ε, ερωτήσεις του κυρίου Πόροβα. Κοιτάξτε, Όντως η περιβαλλοντική συνιστόσα ενσωματώνεται στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, στο εθνικό και κοινοτικό και εκτιμένο. Έχουμε τα επιχειρησιακά προγράμματα σε κάθε χώρα και περιλαμβάνουν πάντοτε ε, στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάντοτε, σε κάθε έργο. Το θέμα είναι ότι την ε, αξιολόγηση αντικτύπου στο περιβάλλον την ε, κάνουν τα κράτη-μέλη και πολύ συχνά αγνοούν ή δεν κατανοούν τη σημασία αυτών των διαδικασιών. Για παράδειγμα, για την ανάπτυξη των μεταφορών, ένα βασικό στοιχείο είναι η επιλογή της εναλλακτικής λύσης και πολύ συχνά αυτό παραγνωρίζεται. Έχουμε δηλαδή την εξή απόφαση, τη απόφαση. Έχουμε αποφασίσει να φτιάξουμε το χύψι αυτοκινητόδρομο ή ε, τη χύψι υδροδρομική σύνδεση. Από εκεί και πέρα, ε, σε ό,τι αφορά στην καταστροφή του περιβάλλοντος, ακόμα και όταν ο αντίκτυπος ε, είναι υπαρκτός, σύμφωνα πάντοτε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά γίνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Και το να αποκατασταθεί το περιβάλλον, αν και όποτε γίνεται, δεν γίνεται στον ίδιο βαθμό, δεν γίνεται στον απαραίτητο βαθμό. Τώρα, ως προς τους διαδρόμους των διευρωπαϊκών δικτύων στο σκέλος των μεταφορών, TNT, πρέπει να σας πω ότι η διάδρομη αυτή είναι εξαιρετικά ακριβή. Ποτέ δεν έχει γίνει στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ουσιαστική ε, ανάλυση οικονομική. Είναι γραμμές που έχουν χαραχθεί πάνω σε ένα χάρτη. Δεν ξέρουμε. Υποπτευόμαστε ότι μπορεί να είναι υπερβολικά ακριβή. Δεν το γνωρίζουμε. Και θέλω να απαντήσω και στο ερώτημα του κυρίου Κράμερ. Ποιες είναι οι επιλογές που υιοθετούμε καθημερινά κάθε φορά που αποφασίζουμε επί ενός συστήματος μεταφοράς. Η απόφαση που παίρνει κανείς σήμερα θα έχει επιπτώσεις στα παιδιά του, στα παιδιά του μετά από 20 ή από 30 χρόνια. Επομένως, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά ε, προσεκτικοί, σόφρονες, επιφυλακτικοί κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Φέρνω το παράδειγμα του διαδρόμου 4. Ε, ε, Είναι ή αυτός που, είναι αυτός που συνδέει το Αμβούργο με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και περνά ε, μέσα από τη Βουλγαρία. Είναι ο διάδρομος που χρησιμοποιείται κατεξοχήν για ε, τις εμπορευματικές μεταφορές. Στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχουμε αυτοκινητόδρομο, ενώ ε, το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ανεπαρκές και δεν μπορεί να ικανοποιήσει ε, τις ε, εμπορευματικές μεταφορές. Εδώ δεν μπορεί καν να μεταφέρει όσους επιβάτες το χρειάζονται. Το χρειάζονται. Από την άλλη πλευρά, για παράδειγμα, η ποδηλασία είναι ανεπτυγμένη στα αστικά κέντρα. Πολλοί ποδηλάτες το, το προτιμούν μέσα στα αστικά κέντρα. Είναι σχεδόν χόμπι. Αλλά δεν έχουμε εθνικό δίκτυο ε, ποδηλατικό στη χώρα μου. Και δεν έχουμε καν την σκέψη να το υλοποιήσουμε και δεν έχει αλλάξει καν η νοοτροπία ότι πράγματι μας χρειάζεται ένα εθνικό ε, δίκτυο πολυδηλατόδρομων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για τις ε, ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Είστε βέβαια πρόσεκτοι να καθίσετε στην αίθουσα μέσα για να παρακολουθήσετε και με τη βοήθεια της επιμελίας την υπόλοιπη συζήτηση. Και πάλι σας ευχαριστώ. So, dann Περνάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο κομμάτι, υποδομές για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ως πρώτο ομιλητή τον κύριο Γιάννου Βίντς, Ευρωπαϊκή Οργάνωση επιβατών θα μας μιλήσει για την προοπτική των επιβατών και τη συνδεσιμότητα με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ και καταρχάς θέλω να ευχαριστώ τον Πρόεδρο και την Γραμματεία της Επιτροπής των Μεταφορών για την ευκαιρία. Με συγχωρείτε, ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, ηρεμία. Δεν είναι καθόλου ευγενικό για τον ομιλητή μας. Uh, ε, ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε εδώ για την προοπτική των επιβατών για τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα διασυνοριακή διασύνδεση. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Ομοσπονδία Επιβατών είναι μια οργάνωση ε, ο ομπρέλα των Ομοσπονδίων Επιβατών, των Ενώσεων Επιβατών. Από το 2002 που ιδρυθήκαμε έχουμε διατηρήσει τις επαφές με, τα, με τις ε, Εθνικές Ομοσπονδίες και ιδιαίτερα το 2007 κάνουμε ε, μία έκθεση κάθε χρόνο για τα ταξίδια χωρίς σύνορα όπου σημειώνουμε προβλήματα ε, διασύνδεσης ή μη μεταξύ κρατών μελών. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την ε, προσχώρηση των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στο χώρο του Σέγγεν υπάρχει πολύ μεγάλη ευκολία στο να διασχίσει κανείς τα σύνορα αν ταξιδεύει οδικός, αν ποδήλατη ή αν περπατεί για να διασχίσει τα σύνορα. Εάν όμως θελήσει να χρησιμοποιήσει τις δημόσιες μεταφορές, τις μαζικές μεταφορές δεν είναι τόσο εύκολο να περάσει τις, ε, τα σύνορα από τη μία χώρα στην άλλη. Μπορώ να σας και τις περιπτώσεις όπου έχει μάλιστα επιδεινωθεί η κατάσταση. Γενικές προϋποθέσεις σε σχέση με, τις, ε, με τα περάσματα αυτά από την προοπτική των επιβατών είναι αντίστοιχα με αυτά που θα πρέπει να περιμένει κανείς γενικά από τις μαζικές ε, μεταφορές, δηλαδή να είναι τακτικά τα δρομολόγια, να ε, ε, τηρείται ένα ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα από τις δύο εμπλεκόμενες χώρες, να πλησιάζει στη μεγαλύτερη πρόσταση, κοντινή στα σύνορα πόλη. να είναι τα τιμολόγια ε, ναι, συγκρίσιμα και επίσης να γίνεται απρόσκοπτα η μετάβαση από το ένα σημείο στο άλλο πέραν των συνόρων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά δυστυχώς σε σχέση με το ιδεό δεν συστηρούμε πολύ. Έχουμε λοιπόν αποστάσεις χαρακτηριστικές από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι οποίες σημειώνουν πολύ περιορισμένες υπηρεσίες Παραδείγματα βλέπετε εδώ από την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης με δύο, τρία, άντε και το πολύ πέντε δρομολόγια πέραν των συνόρων χρήσιμα σχεδόν καθόλου για μεταφορές πέραν των συνόρων. Επίσης ιδιαίτερα σοβαρό θέμα είναι αυτό της τιμολόγησης των υπερσυνοριακών ταξιδιών αυτό το πίνακα νομίζω θα τον γνωρίζετε, κύριε Πάινα, γιατί και εγώ από την ίδια περιοχή είμαι. Βλέπουμε λοιπόν ότι αν θέλουμε να ταξιδέψουμε 30 χιλιόμετρα μέσα στην ε, Ουγγαρία μας κοστίζει μόνο λίγα ευρώ. Ο δε φοιτητής, συνταξιούχος ε, και λοιπές ομάδες πληρώνει και τα μισά ακόμη αυτού του χαμηλού τιμήματος. Αντίστοιχες τιμές βλέπουμε και στην Ρουμανία μέχρι και φθηνότερες. Αλλά εάν θέλει κανείς να διασχίσει τα ολίγα χιλιόμετρα μεταξύ των δύο παραμεθωρίων πόλεων, δεν υπάρχουν καταρχάς ειδικά τιμολόγια και γενικά η τιμολόγηση είναι έως και δεκαπλάσια σε σχέση με μεγαλύτερες ακόμη διαδρομές. Άρα είναι άχρηστο ουσιαστικά αυτές τις συνδέσεις μεταφορά δηλαδή από τη μια μεριά στην άλλη ε, των συνόρων. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τη δική μου δε, ιδιαίτερη πατρίδα, αντίστοιχε αποκλήσει στην τιμολόγηση βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, λυπηρό βλέπουμε το ότι σε πολλές περιπτώσεις οι διασυνδέσει, η κατάσταση επιδεινώθηκε από την ένταξη των εμπλεκομένων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στον χώρο του Σέγγεν. Συγκρίσει συγκριτικά λίγες είναι οι περιπτώσεις που παρουσιάζουν βελτίωση και θεωρούνται καλά παραδείγματα. Από αυτά όμως θα ήθελα σύντομα να τοποθετηθώ προς τη διασύνδεση Αυστρίας, Ουγγαρίας και Σλοβακίας περί τη Βιέννη, στην ευρύτερη περιοχή της Βιέννης, που αποτελεί ένα αρκετά καλό παράδειγμα. Γιατί, γιατί η τιμολόγηση, το χρονοδιάγραμμα και η ε, ολοκληρωμένη προσφορά των υπηρεσιών είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και θα ήθελα επίσης να αφαιρθώ και στην διασυνοριακή γραμμή μεταξύ Σλοβενίας-Ουγγαρίας που έχει πλήρως χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα βέβαια υπάρχει περιθώριο για βελτίωση, αλλά εν γέννη βλέπουμε ότι δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Είναι πολύ καλύτερα από τις αντίστοιχε και συγκρίσιμε σιδηροδρομικές γραμμές σε, άλλες, σε άλλα σημεία της περιοχής. Ε, για να ολοκληρώσω λοιπόν με τα συμπεράσματα, οι περιφερειακές υπηρεσίες εκατέρωθεν των συνόρων πρέπει να προσφέρονται κατά τρόπο συντονισμένο. Τα ε, εσωτερικά τιμολόγια, δηλαδή ουσιαστικά οι επιδοτήσεις προσφέρει ένα κράτος στην τιμολόγηση θα πρέπει να ε, καλύπτουν και την ε, διαδρομή για μετά τα σύνορα, όχι μόνο μέχρι την τελευταία, ε, τον τελευταίο σταθμό πριν τα σύνορα. Η χρηματοδότηση θα πρέπει να υπάρχει. Αν υπάρχει δε χρηματοδότηση υποδομών από ευρωπαϊκά κονδύλια, πρέπει αυτή να αφιερώνεται το μόνο στις υποδομές, αλλά και στην ε, στις υπηρεσίες, ιδιαίτερα για την ε, πρώτη περίοδο, γιατί διαφορετικά τα χρήματα που θα δοθούν στις υποδομές, εάν δεν στηρίζονται και από αντίστοιχε υπηρεσίες, θα είναι πεταμένα από το παράθυμα. Παράθυρο. Έχουν ε, ιδιαίτερα ισχυρού δεσμού οι χώρε αυτέ Κεντρική Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπη παραδοσιακά μεταξύ του και θα ήταν τεράστιο πλεονέκτημα να υποστηριχθούν οι μεταφορές αυτές. Ευχαριστώ και μπορείτε την έκθεσή μα να την κατεβάσετε και από την έκθεσή μα. Ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Κάτριν Όπστ ε, από τους εσωτερικού λιμένες της Ευρώπη για να μας μιλήσει για τις εσωτερικέ πλωτέ οδούς, τις υποδομές ε, και τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, ε, βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή την ακρόαση Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εσωτερικών Λιμένων. Μέλη μας είναι 200 εσωτερικοί λιμένες σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα κλασικό εσωτερικό λιμάνι Μπορείτε να δείτε τη σύνδεση, τη γερσαία και τη σιδηροδρομική και βλέπετε και όλες τις βιομηχανίες που εγκαθίστανται σε ένα λιμένα γιατί βεβαίως εξαρτώνται από την καλή σύνδεση. Οι εσωτερικοί λιμένες διαδραματίζουν διάφορους ρόλους, αποτελούν κόμβους σε αυτό το δίκτυο και συνδέουν τις θαλάσσιες μεταφορές με τις σιδηροδρομικές μεταφορές θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές και σε μικρότερες αποστάσεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αποτελούν μια πλατφόρμα για την περιφερειακή οικονομία. Μπορούμε να μιλάμε για μικρές εταιρείες ή για μεγάλες εταιρείες, σαν τη Volkswagen, που χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους μεταφοράς στο λιμένα των ε, Βρυξελών. Υπάρχει ένας από τους μεγαλύτερους αλευρόμιλους στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να είναι κοντά όλα τα είδη μεταφορών. Αυτές, αυτά είναι τα προαπαιτούμενα για να μπορέσουν να διαδραματίσουν οι λιμένες αυτό το ρόλο και να υπηρετήσουν την οικονομία και την περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να, υπάρχουν, να υπάρχει σύνδεση με όλες, ε, όλα τα μεταφορικά μέσα, με εσωτερικούς ε, ε, ε, ε ποταμούς, με τις σιδηροδρομικές μεταφορές ή με οδικές μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή άρχισε να ασχολείται με το Δούναβι με έναν τρόπο περισσότερο συνεκτικό. Βλέπετε εδώ η σύνδεση Ρότερνταμ-Κωνσταντσα. Είναι σχετικά περιορισμένες οι συγκοινωνίες που χρησιμοποιούν, τα συγκοινωνιακά μέσα που χρησιμοποιούν τον Δούναβι. Βλέπετε τις ε, χώρες που διασχίζει. Η κήτη του ποταμού έχει χαλίκια μετακινείται όμως συχνά και για το λόγο αυτό χρειάζεται διαρκή συντήρηση. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες κατά μήκος του Δανούβιου, ε, Δούναβη που δεν έκαναν την αναγκαία συντήρηση. Όταν είναι χαμηλά τα επίπεδα του νερού σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να φορτώσει τόσο πολύ εμπόρευμα και πράγμα που σημαίνει μείωση των κερδών. Αν το επίπεδο περάσει στα δύο μέτρα τότε παρουσιάζεται ένα έλλειμμα. Τα πλαίσια της στρατηγικής για τον Δούναβι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε, αναπτύχθηκε πρόσφατα ένα σχέδιο αποκατάστασης και εξυγίανσης της περιοχής. Εδώ μπορείτε να δείτε τα σημεία που απαιτείται παρέμβαση. Ίσως σας τρομάξει αυτό. 85 εκατομμύρια ευρώ θα ήταν αρκετά για να φτάσουμε στα ε, συνιστόμενα επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών. Και χρειάζονται βεβαίως άλλα 8 εκατομμύρια για τη συντήρηση του συστήματος. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν και στις διάφορες επιτροπές και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι μάλλον λίγα αυτά τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να προσφέρει κάποια οικονομική στήριξη ως τομέας ζητήσαμε από τους υπουργούς να υποστηρίξουν αυτό το έργο και πραγματικά περιμένουμε να υπάρξουν συμφωνίες του Συμβουλίου που θα υποστηρίξουν αυτό το έργο και θα το προωθήσουν έτσι ώστε να είναι πλωτός ο Ντούναβης και να αποδίδει αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο είναι ο κύριος Μοζότσι. Πρόκειται για τον πρόεδρο της ε, Ένωσης Συντηροδρόμων. Εκπροσωπεί την ε, ε, έποψη των κεντροανατολικών ευρωπαϊκών κρατών σε σχέση με τους σιδηροδρόμους και τις υποδομές του. Παρακαλώ. Sorry. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να παραστώ σε αυτή την ακρόαση και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω για ε, ε τον τομέα αυτό. Την περασμένη εβδομάδα οργανώσαμε μια διάσκεψη στη Βουδαπέστη και αποφασίσαμε να διερευνήσουμε τα προβλήματα και να βρούμε λύσεις η κίνηση η σιδηροδρομική για τις εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να αριθμιστεί σωστά και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν στους κανονισμούς και να ανοίξει η αγορά στον ανταγωνισμό Στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη υπάρχουν και άλλα προβλήματα, όχι σημαντικά για τα 15 κράτη-μέλη, τα παλαιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε λοιπόν αυτή, αυτό το τρένο. Η εικόνα αυτή πάρθηκε κατά την ε, τελετή που είχε οργανώσει η Ουγγροαυστριακή οι που αποκάλυψαν ένα τρένο για την ε, επέτειο της, την 25η του αποκαλούμενου Πανευρωπαϊκού Πικνίκ τον Αύγουστο του 1989 όταν για πρώτη φορά άνοιξε το σιδηρούν παραπέτασμα κοντά στο Σοπρόν το οποίο σιδηρούν παραπέτασμα κάποτε χώριζε την Ευρώπη ε, στα δύο. Μάλιστα, ο κύριος Ολίβιε Ονίδη μας έστειλε ένα μήνυμα με τηλεδιάσκεψη όπου έλεγε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα να χρησιμοποιήσουμε σιδερένιες, σιδηροδρομικές ράγες, όχι για να χωρίσουμε, αλλά για να ε, συνδέσουμε την Ευρώπη και να φτιάξουμε ένα ενιαίο ε, δίκτυο ε, σιδηροδρομικών μεταφορών. Ελπίζω η Ουγγαρία και οι άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να έχουν ρόλο καθοριστικό για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και μας είπε μάλιστα ότι η Επιτροπή με χαρά θα συνεργαστεί για να, για επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ποιες είναι όμως οι προκλήσεις για τις συνδρομικές εταιρείες που ασχολούνται με τις εμπορευματικές μεταφορές. Ε, οι πρώτες τρεις προκλήσεις είναι πολύ σημαντικές, γιατί υπάρχει ανταγωνισμός με τις οδητικές μεταφορές και τις πλωτές οδούς. Η τέταρτη πρόκληση είναι η πολιτική ε, πρόκληση και αυτή είναι ευθύνη των κρατών μελών. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την ε, κίνηση του σιδηροδρόμου, να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η σιδηροδρομική σύνδεση και να ενσωματώσουν την εθνική νομοθεσία. τι περιμένουν οι πελάτες, οι χρήστες από τους σιδηροδρόμους, ανταγωνιστικές τιμές με στήριση των χρονοδιαγραμμάτων και ασφάλεια. Αυτά είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες. Όμως ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τα τέλη είναι εξαιρετικά υψηλά, η υπηρεσία που προσφέρεται είναι κακή και ο χρόνος μετάβασης ταξιδιού είναι πολύ μεγάλος. Έχουμε μη συντονισμένες ιδιοκτησίες των γραμμών, αν θέλετε, στις διάφορες γειτονικές χώρες, διαφορετικούς περιορισμούς, ε, πάρα ε, πολύ μεγάλους χρόνους αναμονής στα σύνορα ή από την μία διοικητική επαρχία στην άλλη. Πρέπει να έχουμε βελτιωμένη αποδοτικότητα της ε, διαχείρισης της ε, κίνησης μέσω σειροδρόμου και των εμπορευματικών μεταφορών. Η λύση λοιπόν είναι στο Rail Freight Corridors, ε, στο να έχουμε διαδρόμους σιδηροδρομικούς για τις εμπορευματικές μεταφορές. Πρέπει να λύνονται τα προβλήματα των πελατών, των καταναλωτών. Τα κανονιστικά μέτρα για τους διαδρόμους είναι τα πιο σημαντικά. Ε, χάρηκα όταν διάβασα αυτούς τους σχετικούς κανονισμούς για πρώτη φορά, γιατί κατάλαβα ότι μόνο με ευρωπαϊκό συντανισμό μπορούν τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τη συντροδρομική εμπορευματική μεταφορά και την κίνηση σε αυτά τα δίκτυα. Πολύ συχνά οι φορείς εκμετάλλευσης των σιδηροδρόμων δεν συμφωνούν για τους περιορισμούς, δεν δίνουν σωστά στοιχεία και πληροφορίες έγκαιρα, δεν προσφέρουν εναλλακτικέ διαδρομές. Μια κοινή ε, πολιτική για τα τέλη χρήσης της υποδομής μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχία του σχεδίου μας. Η διαλειτουργικότητα, όλα αυτά τα πρότυπα ε, στα οποία πρέπει όλοι να συμμορφωθούν ή ε, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πελωτών. Πελατών, με Βλέπετε εδώ τις βασικές παραμέτρους των διαδρόμων. Σε ορισμένες χώρες αυτά είναι όνειρα και σε άλλες χώρες είναι πραγματικότητα. Έχουμε για παράδειγμα μια γέφυρα σιδηροδρομική μεταξύ δύο χωρών, αλλά οι γραμμές που συνδέουν δεν επιτρέπουν απρόσκοπτη ε, κίνηση λόγω χαμηλής ταχύτητας ή άλλων περιορισμών. Εδώ βλέπετε το ε, πυρήνα, τα βασικά δίκτυα διαδρόμων τα διευρωπαϊκά. Έχουμε τους εννέα διαδρόμους και η περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενδιαφέρεται για τους τέσσερις από τους εννέα. Η Τουρκία, ε, η οποία δεν είναι κράτος μέλος, είναι πολύ σημαντικός πελάτης και χρήστης των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Ε, όλοι θέλουν να έχουν καλές επιχειρηματικές σχέσεις με την Τουρκία και αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Ε, λόγω των προβλημάτων τα οποία τόνισα, ο σιδηρόδρομος δεν είναι σε πολύ ανταγωνιστική θέση σήμερα στην κεντρική ε, Ευρώπη, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, γιατί υπάρχουν πλοία μεταξύ Ιταλία και Ελλάδας, Ιταλίας Τουρκία που ε, ε, μεταφέρουν τα εμπορεύματα χωρί πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να αρθούν όλα αυτά τα εμπόδια που οδηγούν σε ε, κυκλοφοριακή συμφόρηση στι υδροδρομικέ εμπορευματικές μεταφορές. αυτά τα εμπόδια είναι που στηρίζουν τις πλωτές οδούς και θα πρέπει επίσης να πούμε ότι υπάρχουν παράμετροι σε σχέση με τις ε, υποδομές που συμβάλλουν στο πρόβλημα. Έχουμε χρόνους αναμονής που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, άρα ψηλότερο κόστος. Δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών ε, μεταξύ ε, των διαφόρων φορέων εκμετάλλευσης. Δεν υπάρχει συντονισμός, κοινός σχεδιασμός κ.ο.κ. Όλα αυτά έχουν συνέπειες. Γιατί πολύ συχνά μέχρι ότου φτάσει το τρένο στο λιμάνι θα έχει ήδη φύγει το πλοίο και το καθεξής. Για να έχουμε πολυτροπικό τρόπο μεταφοράς λοιπόν, πολυτροπικές μεταφορές πρέπει να έχουμε καλύτερα, καλύτερο συντονισμό. Χρειάζεται ευρωπαϊκό συντονισμός και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα μέσα του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη ή το Ταμείο Συνοχής Πιστεύω ότι η ανάπτυξη πολυτροπικών τερματικών σταθμών είναι εξαιρετικά σημαντική και θα πρέπει να στηριχθεί η σιδηροδρομική σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτέ ήταν λοιπόν οι παρουσιάσει από τους ομιλητές μας. Παρακαλώ, ερωτήσεις και απαντήσεις. Κύριο Σερτού, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερω για τι πολύ ενδιαφέρουσε παρουσιάσει Για την κυρία Όπστ έχω μια ερώτηση. 85 εκατομμύρια ευρώ που θα χρειαστούν εν τέλει. για να καταστεί τόσο ο Δούναβης. Από πού τα βγάζετε τα 85 εκατομμύρια και επίσης, μια άλλη ερώτηση, το κομμάτι ε, που εξαιρείται μεταξύ Φάσεν και Φερσόφεν ή μάλλον το πω διαφορετικά, είναι ρεαλιστικό να λέμε ότι ο Δούναβης όπως έχει τώρα η κατάσταση μπορεί να γίνει πλωτός όπως και ο Ρήνος και να απελευθερωθεί στις μεταφορές όπως ο Ρήνος. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές μεταξύ κρατών και διορισμένων κρατών. Ο Πρόεδρος, ε, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Αν όχι, έχω εγώ ερώτηση για τα δικαιώματα των επιβατών καταρχάς. Οι συνδέσεις ανατολικά της Βιέννης προς τρία κράτη, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, με υπερσυνοριακές ε, διαδρομές και ίδια τιμολόγια. Αυτό όμως το βλέπουμε να συμβαίνει αλλού. Με κάποιο τρόπο το καταφέρατε λοιπόν εσείς. Οι άλλοι μα λένε έχουν προβλήματα. Γιατί λοιπόν μπορείτε μεταξύ Σλοβακία, Ουγγαρία και Αυστρία να έχετε τα ίδια τιμολόγια και υπερσυνοριακέ ε, διαδρομέ και δεν το καταφέρουν τα άλλα κράτη. Αυτό πρώτον, πολύ σημαντικό. Δεύτερον, διάβαση των σύνορων, cross-border. Μπορώ να σα δώσω πολλά παραδείγματα, αλλά θα σα αναφέρω το SELP ARSH, 8 χιλιόμετρα όλα και όλα, που ήταν χωρισμένα από το σιδηρούν παραπέτασμα στο παρελθόν, πολύ περιορισμένη η έκταση. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να γίνει η διασύνδεση και ετοιμολόγια καλά θα μπορούσαμε να έχουμε κτλ. Αλλά φαίνεται ότι κανείς δεν σκέφτεται να πάει το τρένο μέχρι την, τον επόμενο σιδηροδρομικό κόμβο ή μέχρι το προηγούμενο να γίνει αντίστροφα η διασύνδεση και πάντως με το ίδιο τιμολόγιο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως. Το Βερολίνο Στετίν με την ε, ε, πρώτη κατασκευή της σιδηροδρομικής διασύνδεσης ήταν πολύ υψηλό το τιμολόγιο αρχικά πρέπει να σας πω ήταν πολύ ακριβό για την Πολωνία βασικά και έτσι πήγαιναν άδεια τα τρένα Εν τω μεταξύ όμως συνεννοήθηκε το Βερολίνο με το, κράτος, με το κρατήριο του Βαρδεμβούργου ώστε να πέσει το εισιτήριο στα 10 ευρώ αφενός αφετέρου δε να είναι η τιμολόγηση αντίστοιχη είτε έρχεται κανείς από το Βερολίνο είτε έρχεται από το Στετίν. Ε τώρα είναι γεμάτα τα τρένα και μπόρεσαν να γεμίσουν όχι χάρη στην υψηλότερη τιμολόγηση, αλλά στο χαμηλότερο εισιτήριο. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Δεν έχει νόημα να μένει έχουμε επιβάτε να πηγαίνουν τα τρένα με υψηλέ τιμέ, αλλά να είναι άδεια. Ε, Επίση για τα σόπον, θυμόμαστε πολύ καλά το 25ο εκείνο πανευρωπαϊκό πικνίκ. Υπάρχει μια διασύνδεση από την Βιέννη, των Σόπων στο Ζάγκρεπ, στη Λουμπλιάνα και το Κοπα... Ε, κάποιες από τις γραμμές αυτές ή κάποια από τα κομμάτια της γραμμής ε, μπορεί να χρειάζονται ακόμα και ράγες ή απλώς ηλεκτροδότηση. Αλλά πάντως υπάρχει αυτή η γραμμή. Και αντίστοιχα έχουμε το, το, βαλτικό διάδρομο με, τον, ε, με, το, με τη σύρεγγα των Άλπαιων και του Σέβεριν μετά. Ερωτώ λοιπόν, γιατί να μην ξεκινάτε με τη βασική δουλειά και ας μείνει για αργότερα ενδεχομένω η σύρεγγα από το να μην γίνεται τίποτα. Γιατί θα ήταν εύκολα, θα ήταν εύκολο να μειωθεί κατά 6-7 ώρες το ταξίδι από τη Βιέννη μέχρι το Ζάγκρεπ. Μόνο αν είχατε κάνει τα, τα, τα, τα κομμάτια της διαδρομής που είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Κοιτάω γύρω μου, αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, σας δίνω το λόγο και να απαντήσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Δύο ερωτήσεις απευθύνθηκαν σε μένα. Η μία αφορούσε 85 εκατομμύρια απόθεν τα βλέπουμε εμείς. Πρόκειται για μια μελέτη που έγινε στο πλαίσιο της στρατηγικής ε, του χώρου του Δούναβή, δηλαδή από τη γραμματεία της ε, στρατηγικής για το Δούναβη και σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα κράτη, τα οποία έπρεπε να μας πούνε πόσο περίπου κόστος υπολόγιζε το καθένα για το δικό του κομμάτι, άρα έχουν συνεργαστεί και τα κράτη. Το master plan θα συζητηθεί από ό,τι ξέρω αύριο στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Άρα, άπαξ και συζητηθούν και τα ε, αριθμητικά που σας ανέφερα, νομίζω επιβεβαιώνονται. Επίσης, αν μπορεί να γίνει μια εξομοίωση μεταξύ των δυνατοτήτων του Δούναβη και αυτών του Ρήνου για, πλω... για χρήση ως πλωτής οδού. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό λίγο ρίχνει τον Δούναβη, γιατί ο Ρήνος ξεκίνησε και λόγω της παραδοσιακής ανάπτυξης των βιομηχα... της βιομηχανικής παραγωγής, της όχθες του και έχει αναπτυχθεί. Ο Δούναβης δεν έχει το ίδιο, το ίδιο ιστορικό, δεν έχει την ίδια βιομηχανική παραγωγή αλλά έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, εγώ δεν θα έλεγα να κάνουμε το Δούναβι κάτι σαν αλλά να αναπτύξουμε το υφιστάμενο δυναμικό του Δούναβη. Ο Δούναβι, σε παραδείγματι, έχει στη βιομάζα τεράστιο δυναμικό. Αυτό πρέπει να το ψάξουμε. Πείτε. Παρακαλώ εσείς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος Βίντσε. Αναφερθήκατε στο κομμάτι Βιέννη, Σόμπρον, Ζάγκρε, Μπλουμπλιάνα. Έχουμε δύο κομμάτια στη σιδηροδρομική αυτή γραμμή που δεν έχουν λειτουργηθεί ακόμη μέσα στην Ουγγαρία. Και δεν έχουμε και διπλές γραμμές. Ράγκες δηλαδή. Η Ουγγαρία έχει επιλέξει στρατηγική να ηλεκτροδοτήσει συγκεκριμένες γραμμές. Για το Βιέννη Γκράτς και για, τις, ε, το κομμάτι Άλπης Αδριατική είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα. γιατί ήδη βλέπουμε ότι το κομμάτι που αφορά το Σενκοντάρ έχει εξυγχρονιστεί πάει πολύ γρήγορα το τρένο μέχρι και 160 χιλιόμετρα, έχει σύστημα EMTS και βλέπω τώρα σε σχέση με το τέλος χρήσης των, της ράγας, των στριοδρόμων δηλαδή, στο Ζέμερινγκ, ότι υπάρχει δυναμικό γι' αυτό ίσως υπάρχει ανάγκη να ηλεκτροδοτηθεί το κομμάτι μεταξύ Γκράτς και Ουγγρικών συνόρων. Αυτό είναι το έλλειμμα. Εδώ χρειάζεται συμφωνία μεταξύ των δύο κρατών ή ευρωπαϊκά κονδύλια για τις υποδομές αυτές. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κύριε Βίντσε, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον κύριο Κράμερ. Πράγματι, υπάρχουν καλά παραδείγματα στην περιοχή της Βιέννης και την ευρύτερη περιοχή. Ε, θα πρέπει να αντιγραφούν, να εμπνευστούμε από αυτά και να δούμε ε, σε ποια σημεία οι επιδόσεις μας είναι ε, πιο αδύναμες. Και αν δούμε την περιοχή της, Βιέννας, της Βιέννης, ε, το κοντράστι, η αντίθεση, είναι πολύ σοκαριστικό. Γιατί οι μεταφορές από Αυστρία στην Ουγγαρία και από Αυστρία Σλοβακία, Σλοβακία έχουν βελτιωθεί ιδιαίτερως. Έχουμε ένα ενιαίο σύστημα αυτή τη στιγμή. Όμως, μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβακίας, στην ίδια περιοχή Έχουν κλείσει όλες οι συνδέσεις μεταφοράς επιβατών ή μέσω σιδηροδρομικής ε, σύνδεσης και το καθεξής. Δεν το λέω για να πω ότι δεν υπάρχει δυναμικό στο Νότο. Φυσικά και υπάρχει. Ωστόσο, οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, ο κόσμος αλλά και οι κυβερνήσεις δεν έχουν αυτή την οτροπία. πρημοδότησης των δημοσίων μεταφορών ή συγκοινωνιών έτσι ώστε να έχουν αυτές τη θέση που τους αξίζει. Το είπαμε σήμερα, το συζητήσαμε. Πολλοί στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θεωρούν ότι τα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι εναλλακτική τύπου Β σε σχέση με την Α εναλλακτική που θα ήταν να έχει ο καθένας το ιδιωτικό του αυτοκίνητο. Ενώ στην περίπτωση της Βιέννης ή του Βερολίνου η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται και βελτιώνεται δραματικά. Είναι δηλαδή και θέμα αντίληψης. Ελπίζω λοιπόν όταν μια χώρα στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη έχει τέτοιο πρόβλημα να εμπνέεται από την άμεση γειτονική της χώρα που ανήκει στην παλιά εντός εισαγωγικών Δυτική Ευρώπη για να ε, λύνει τα προβλήματά της και να αλλάζει η νοοτροπία προς το καλύτερο. Σίγουρα οι υποδομές είναι εξαιρετικά ακριβές και πρέπει να αξιοποιούνται. Πράγματι δεν υπάρχει λόγος να γίνονται υποδομές χωρίς να χρησιμοποιούνται. Έχουμε διασυνοριακές πλέον υποδομές στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ίσως όχι τόσο καλές όσο στη Δυτική Ευρώπη, αλλά εν πάση κάθε κονδύλιο που υπάρχει πρέπει να αξιοποιείται για να ε, βελτιωθούν αυτές οι υποδομές ε, και να γίνει το καλύτερο δυνατό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τις εννέα λοιπόν παρουσιάσεις. Έγινε μια πολύ ζωντανή συζήτηση, την οποία παρακολούσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα παρακαλώ την Έλληνα Πίντο εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο, αλλά θέλω να προσθέσω το εξή, αν σα κατάλαβα καλά. Ορίζονται επίτηδε ορισμένα τιμολόγια πολύ υψηλά, ώστε να μην χρησιμοποιείται ένα κομμάτι διαδρομής προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα ενός φερρυπίν τούνελ μια σύραγα που θα χτιστεί σε 10 χρόνια. καταλαβαίνω καλά ότι δηλαδή δεν ηλεκτροδοτείται ένα κομμάτι του δικτύου προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστικό για κάτι που βρίσκεται μόνο σε προοπτική. Θα μας το επιβεβαιώσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως κάνουμε και ένα παραλυσμό σε σχέση με το Σεφερμέ και την, ε, την προώθηση εναλλακτικών ε, διαβάσεων. Ο πρόεδρος, ο κύριος Μοσόσκι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Το έχω μελετήσει αυτό σε πολλά κράτη. Είναι προφανές ότι προωθούνται συγκεκριμένες διάδρομες και εάν πρόκειται να έρθουν νέα τρένα, δηλαδή χρειάζονται υποδομές πιο προηγμένες ε, κτλ, τότε ορίζεται πιο υψηλό τίμημα. Το ίδιο με το Σέμεριν στην Αυστρία, που επειδή δεν έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, έχει χαμηλότερες τιμές. Αν θέλει κανείς να μεταφέρει κάτι μεταξύ του Σενκοτάρ και της ε, Αυστρίας, υπάρχει αυτή αυτός ο σύρμος. Και αν κανείς δεν χρησιμοποιεί τις ηλεκτροδοτούμενες ε, γραμμές, είναι πιο φθηνά τα πράγματα. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Δηλαδή, τώρα στη Γερμανία, ξέρετε που μειώνεται το διόδι, τα διόδια, μειώνονται τα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα φορτηγά, με το επιχείρημα ότι μάλλον αυξάνονται τα διόδια για τα φορτηγά με το επιχείρημα ότι έχουν πέσει τα τιμήματα των υποδομών και άρα χρειάζεται χρήμα. Έχετε το λόγο κυρία Πίντο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Ε, προσωπώ την αρμόδια υπηρεσία που ασχολείται με τα δικτυακτά δίκτυα μεταφορών. Η συζήτηση εδώ υπήρξε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα Ακούσαμε πάρα πολλά παραδείγματα σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι το να είναι καλές αυτές οι διασυνδέσεις. Ξέρουμε ότι η κατάσταση στις ε, χώρες που βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη. Θα ήθελα να πω ότι η Επιτροπή βεβαίως έχει γνώση του προβλήματος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξουν διακρατικές συνδέσεις. Οι υποδομές είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μια έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών ή ε, ενδεχομένως υπάρχει ελλειπής ε, ε, διάθεση από πλευράς των κυβερνήσεων. Συνεπώς, το νέο μέσο για το, το είναι σημαντικό, αλλά και οι διάδρομοι, αλλά και οι Ευρωπαίοι συντονιστές, όπως αναφέρθηκαν εδώ. Θα ήθελα να θυμίσω, μιλώντας για τα διδικαϊκά δίκτυα, ότι τα πλέον σημαντικά για μας είναι τα διακρατικά. Εδώ μιλάμε για διαδρόμους και προβλέπουμε ότι υπάρχουν και θέματα διαλειτουργικότητας όπως τα αναφέρουμε. Αυτό είναι ένα θέμα που επίσης θα πρέπει να μας απασχολήσει. Η αριθμή είναι πάρα πολύ σημαντική, καθώς και το θέμα της χρηματοδότησης. Το 50% της χρηματοδότησης θα πάει σε δρόμους, στο δικό δίκτυο. Για το λόγο αυτό καταβάλλεται μια προσπάθεια να εστιαστεί η προσοχή στους συνδυοδρόμους αλλά και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Ένα άλλο θέμα αφορά τη, διασυνδέσεις που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητήθηκε στο τελευταίο πάνελ. Οι εσωτερικοί λιμένες είναι σημαντικοί αλλά δεν μπορούν να υπάρξουν ε, όταν ε, λείπει το δικτυοκό ή σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι διασυνδέσεις. Ορισμένοι ομιλητές αναφέρθηκαν ότι δεν θα πρέπει να μιλάμε μόνο για την διασύνδεση όταν μιλάμε για τις δικρατικές υποδομές. Θα πρέπει να τα δούμε ως κάτι συμπληρωματικό. Και αυτό είναι κάτι που εξάλλου ανέφερε, ανέφεραν οι Πολωνοί για την Καρπαθία Οδό. Εκεί προσπαθούν να ανασυμπληρώσουν διάφορες χρηματοδοτικές πηγές και θεωρούμε ότι η προσέγγιση αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Το ίδιο γίνεται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν μιλάμε για ταμεία συνοχής και τα κονδύλια από το Ιντερέγκακ. είναι σημαντικά και υπάρχει συνεργασία μεταξύ των δύο τομέων. Εντέθησαν ορισμένα θέματα σχετικά με το πόσες περιφέρειες εμπλέκονται εδώ σε αυτούς τους διαδρόμους. Θα ήθελα να επανέλθω στο έργο των Ευρωπαίων συντονιστών. Εκεί έπαιξαν κάποιο ρόλο οι περιφέρειες και εμείς προσπαθούμε να στείλουμε αυτό το μήνυμα που ακούστηκε σήμερα. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα έργα που υπάρχουν, πιθανότητες, υπάρχουν πιθανότητες να πάρουν χρηματοδότησες και ποια ενδεχομένως θα πρέπει να στραφούν προς τα κανονικά διαθροτικά ταμεία. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ χωρών βελών ή μεταξύ περιφερειών. Αυτό είναι κάτι που πραγματικά προσπαθούμε να προωθήσουμε προς τους συντονιστές. Ακούσαμε ορισμένες ιστορίες επιτυχίας Βεβαίως υπάρχουν ορισμένα θέματα, αλλά όπως είπατε και εσείς η συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Το πώς θα χρηματοδοτήσουμε την πλευσιμότητα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. και την χάνει της στήριξης της Επιτροπής και των Ευρωπαίων Συντονιστών. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα προβλήματα με τις χώρες ε, της προβεσβασιμότητας των χωρών της Βαλτικής και την έλλειψη διασυνδέσεων είναι ένα σοβαρό θέμα. Αυτό είναι ένα από τα πιο βασικά έργα. Θα ήθελα να τελειώσω την παρέμβασή μου λέγοντας ότι έχουμε πλήρες πληροφορίες εδώ όπως ξέρετε, έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας, αλλά υπάρχει ένα πλαίσιο και θα πρέπει να το εφαρμόσουμε. Να το εφαρμόσουμε όμως μαζί, όπως τονίστηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, κατελεκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ όλους τους εδώ παρισταμένους τελευταία μας συνεδρίαση για φέτος. Γι' αυτό είχαμε και μια πολύ σύντομη δεξίωση το μεσημέρι. Ε, πρέπει να αποχαιρετήσω όμως δύο συναδέλφους, την Κριστίνα Ρέτκλιφτ, η οποία φεύγει όχι μόνο λόγω μητρότητας, αλλά μετά θα πάει και στο Policy Department. Κοντά μας θα είναι πάλι. Είναι σχετικό. Δεν θα είναι όμως πια στη γραμματεία της Επιτροπής των Μεταφέρων. Της ευχόμαστε κάθε καλό για το μέλλον και για τους δυο σας, για να μην πω και για τους τρεις σας πια. Και ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία και την υποστήριξη στην Επιτροπή μας. Η δεύτερη που θα μας Ο δεύτερος που θα μας εγκαταλείψει είναι εδώ, ο εκδεξιών μου, Μίχαλ Κοτσικόφσκι, ο οποίος φεύγει από τις μεταφορές και πάει στη Γεωργία. Τον ευχαριστούμε τον Μιχαήλ θερμά για την υποστήριξη, για τη συνεργασία. Και πολύ πολύ κουράγιο για την Επιτροπή Γεωργίας. Und damit wäre die Sitzung... Και ως εκ τούτου κυρίσω το πέρα στις τελευταίες αυτής συνεδριάσεις για το 2014. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, καλές γιορτές και πολύ καλό νέο έτος.